Sí. Is dear. We are going, we are going to start. Θα ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Όπως βλέπετε δεν είμαι ο Μπούζεκ. Είμαι ο Μαρτίνες, είμαι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος υπεύθυνο για τις σχέσεις με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ο κύριος Μπούζεκ μου ζήτησε να συμπροεδρεύσω με τον φίλο εδώ, τον Περ τον πρόεδρο του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσω στην ισπανική γλώσσα. Ανάμεσα στα άλλα θυμίζω ότι είμαι υπεύθυνο και για την πολυγλωσία στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου και θα ήταν προδοσία στις ευθύνε μου να μην χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Συνεπώς, άρχεται η συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Σας ε, καλωσορίζω όλους, σας χαιρετώ και σας θυμίζω αυτό που μου λένε από τη γραμματεία ότι θα πρέπει σιγά σιγά να συμπληρώνετε κάτι έντυπα Δηλαδή όσοι θέλουν να μιλήσουν πρέπει να ζητούν το λόγο. Και μιλώ για τη ε, συζήτηση με τον Σουηδό Υπουργό Δικαιοσύνη και με τον Επίτροπο κύριο Μπαρό. Αν θέλετε να μιλήσετε παρακαλώ συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο. Και ε, σιγά σιγά το παραδίδεται για να εγγραφείτε στο κατάλογο των ομιλητών ε, για την επόμενη συζήτηση. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τώρα 40 λεπτά παρουσίαση των εκθέσεων των ομάδων εργασία. 1, 2 και 3 που συνεδρίασαν εχθέ. Αλλά δεν βλέπω τον κύριο Λόπε Αγγιλά. που θα πρέπει να παρουσιάσει κανονικά την έκθεση πρώτη πρώτης ομάδας εργασίας και μαζί με τον συνάδελφο Βέστερμπεργκ και για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το χρόνο θα περάσουμε σε άλλη ομάδα. Στην ομάδα εργασία 2 και στον κύριο Ράφσαμ από τη Σουηδική Βουλή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αρχίζουμε από τη δεύτερη ομάδα. Παρακαλώ, πέντε λεπτά μόνο ο καθένας να μιλάτε. Tack så mycket. Jag kan inledningsvis nämna σύντομα θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Θα παρουσιάσω την έκθεση από την ομάδα εργασίας 2. Πάρα πολλοί συνάδελφοι και από το Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια είπαν ότι βασικός στόχος είναι να καταστήσουμε τα νομικά συστήματα συμβατά μεταξύ τους σεβόμενοι πάντα τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις κάθε κράτους μέλους βέβαια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν αντιρρήσεις για την κατάργηση της διαδικασίας εξκουάτουρ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ανάμεσα στις απόψεις που ακούστηκαν τέθηκε το ότι ποικίλει η ποιότητα των διοικητικών αποφάσεων στα διάφορα κράτη-μέλη και τις καθιστά ε, μη συγκρίσιμες πάντα μεταξύ τους. Δεδομένης αυτής λοιπόν της κατάστασης έχει σημασία να υπογραμμίσουμε την μεγάλη σημασία που έχει η λεγόμενη νομική βεβαιότητα η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπάρχουν και διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με το πεδίο του δικαίου στο οποίο αναφέρομαι. Το οικογενειακό δίκαιο σαν παράδειγμα ε, αντιμετωπίζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό στα πλαίσια μιας τέτοιας προσπάθειας οι συνάδελφοι να συζητούν τα θέματα του κοινοτικού δικαίου και να προσπαθούν να δουν ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι το φυσικό επόμενο βήμα για μας θα πρέπει να είναι η κατάργηση της διαδικασίας του εξεκουάτου. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης σας ευχαριστώ για τη συντομία σας. Είστε πολύ φοδολός στη χρήση του χρόνου. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή της πρώτης ομάδας εργασίας που κατέφθασε, ο κύριος Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ. Πρόεδρος τη Επιτροπής Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπείων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω στην ομιλία μου το πνεύμα και το γράμμα της συζήτησης που έγινε χθε που ήταν ενδιαφέρουσα όσο και χρήσιμη στην ομάδα εργασίας ε, στην οποία είμαι εισηγητή. Τίτλος «Οικοδόμηση τη Ευρώπης των πολιτών». χτες το μεσημέρι στην πρώτη μου παρέμβαση και στη συνέχεια στη συζήτηση επέμεινα στη σημασία αυτής της κομβικής κεντρικής ιδέας της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομιμότητας, νομιμοποίησης από τους πολίτες. Είμαστε ευρωβουλευτές και βουλευτές Ευρωπαίοι και εκπροσωπούμε Ευρωπαίους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Οι πολίτες λοιπόν έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε εμάς και στο κοινοβούλιο μας και ελπίζουν και περιμένουν από το Κοινοβούλιο απαντήσεις για να βελτιωθούν οι εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και να κατοχυρωθούν. Επιπλέον, χτες έγινε μια συζήτηση ε, που ασχολήθηκε με τις αρχές αυτές, τις μελέτησε και τόνισε ότι η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε αξίες, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, είναι λοιπόν μια οικοδόμηση που έχει τα θεμελιά της στις συνταγματικές παραδόσεις ε, κάθε κράτους μέλους. Αλλά επίσης τη συγκεντρώνει και της ε, σύγγερνα και μετά από μια ε, παρατεταμένη συζήτηση που έγινε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δέκα χρόνια τελικά μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνθέσει και να καταλήξει σε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή με την ευρωπαϊκή λοιπόν, οικοδόμηση και την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και αυτό που κρυσταλλώνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας που συμπεριλαμβάνει και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, γνωρίζουμε και άλλωστε εκφράστηκε και χθε αυτό ότι υπάρχουν επιφυλάξει από κάποια κράτη-μέλη για το εάν και κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη συνθήκη. Ωστόσο, παραμένει γεγονός ότι είναι από τα τρία βασικά στοιχεία της συνθήκης Λισαβόνας μαζί με την αναθεωρημένη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και ο χάρτης των μελιδών δικαιωμάτων και ε, χαράζει ένα νέο ορίζοντα, ένα νέο κοινό παρονομαστή που συνθέτει, όπως σας είπα, τις συνταγματικές παραδόσεις, τις βελτιώνει και τις εμπλουτίζει, χωρίς όμως να αποδυναμώνει τα δικαιώματα των οποίων απολαμβάνουν πολίτες από την ηθαγένειά τους, ως πολίτες ενός κράτους μέλους. Τι σημαίνει αυτό. Κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που γαθορίζονται και κατοχυρώνονται στο χάρτη δεν έρχονται να υποκαταστήσουν, ούτε να καταργήσουν, ούτε να αντικαταστήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των οποίων απολαμβάνουμε ως ε, πολίτε της χώρας μας, του κράτους μας ο καθένας. Επαναλαμβάνω, τα εμπλουτίζουν και τα πολλαπλασιάζουν. Βεβαίω τα ενημερώνουν κιόλα, τα θεωρούμε, γιατί εξελίσσεται συνταγματικά η Ευρώπη και θεσμικά γιατί έχουμε και δικαιώματα νέας γενιάς εντός εισαγωγικών που δεν έχουν ε, κατοχυρωθεί και αναγνωριστεί στα διάφορα συντάγματα. Γιατί προχωρεί η τεχνολογία, έχουμε ε, ανάπτυξη των επιστημών, της βιογενετικής, η κοινωνία της προφορίας, όλα αυτά είναι νέα δικαιώματα. Και επίση έχουμε τις εγγύησεις της ασφάλειας και της ε, προστασίας ιδιωτικής ζωής. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός αυτό και το πρόγραμμα της Σοκχόλμης, διότι σημαίνει στρατηγική δράση για να οικοδομηθεί αυτός ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που ξεπερνά πλέον το διακυβερνητικό στάδιο ε, το οποίο γνώρισε τα τελευταία δέκα χρόνια και έχουμε πλέον μια ευρωπαϊκή πολιτική που υπάγεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα είναι συνομοθέτης και αποφασιστικός. Οπότε κάτι άλλο που συζητήσαμε χθε, ήταν η συζήτηση για το διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί γίνονται συζητήσεις και στα Εθνικά Κοινοβούλια για κάθε ένα από τους στόχους μας ξεχωριστά. Ας πούμε, για... Ε, τι, γίνεται με την ασφάλεια και πώς αυτή συνδυάζεται με το δικαίωμα του πολίτη να έχει προστατευμένη ιδιωτική ζωή. Έχουμε διατλαντικό διάλογο, ξέρετε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι πρόκληση πάντα στη συζήτηση που είχαμε και μάλιστα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ε, την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών την κυρία Τζάνετ Ναπολιτάνο που είχε έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε συζήτηση πάρα πολύ ζωηρή με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερωτήσεις, απαντήσεις, για να δούμε και να εξασφαλίσουμε αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες και ενδιαφέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προστασία της ιδιωτική σφαίρας το δικαίωμα στην προσωπικότητα του καθενό, το δικαίωμα σε μια ε, ιδιωτική σφαίρα πρόστατευμένη, απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις της, της με άλλους για την ασφάλεια και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο θέμα που μας απασχόλησε. Τα δικαιώματα των προσώπων, τα ατομικά δικαιώματα δηλαδή. Και αυτό το συζητούν και τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι γίνεται με ε, πολίτες που δεν είναι πολίτες της Ένωσης αλλά βρίσκονται στην επικράτεια. Είναι και εκείνοι πρόσωπα που χαίρουν ατομικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων. Είτε είναι ε, νόμιμη η μετανάστευση είτε είναι παράνομη. Οι μετανάστες βρίσκονται ε, μεταξύ μας, είναι, ζουν ανάμεσά μας καλή η καταστολή της παρανομίας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Δεν μπορεί κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στη μετανάστευση και την εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά τελείως διαφορετικά ε, ζητήματα. Δεν είναι το ίδιο μετανάστης, είτε νόμιμος είτε μετανάστης, με ε, ε, ξέρω, πω κακοποιό σε μια χώρα. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ναι, πέντε λεπτά είχατε όμως. Τελειώνω. Έτσι λοιπόν. κατέστησε σαφέ ότι η θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και η έγκριση του προγράμματο Στοχόλμη δεν θα διευκολύνει τη ζωή μα ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Το αντίθετο, θα είναι πιο δύσκολη η ζωή μα, πιο πολλέ και μεγαλύτερε οι απαιτήσει των καιρών. Αυτό είναι χρήσιμο για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μα όμω σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά στι ε, υποχρεώσει που έχουμε και στι προσδοκίε που έχουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτε. Συμπέρασμα. Μετά από δέκα ε, ετών σκληρή δουλειά στα θεσμικά δεν θα κατανοούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες τώρα να αποτύχουμε. Να μην συμφωνήσουμε, να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Θα πρέπει να δοθεί σημαντική όθηση από τα κοινοβούλια μας στον χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσεις που επαναλαμβάνω υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια και όρια των κρατών μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία, τη ποινική δικαιοσύνη, κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη τρομοκρατία, κάθε είδου βία και προστασία των θυμάτων. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα και θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να το εγκρίνουμε στο πρόγραμμα της Οχόλμης. Ελπίζω να είναι πολύ μεγάλη συνένεση και να δοθεί συνέχεια και από τα Εθνικά Κοινοβούλια με το πρόγραμμα δράσης της Στοχόλμης που θα τεθεί σε ισχύ το άλλο εξάμενο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την ανοχή σας. Ε... Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κάρμεν Ερμοσίν που είναι η συγγήτρια της τρίτης ομάδας πρέπει να σου πω ότι νιώθω μεγάλη συζήτηση. Αν μας είχε πει κάποιος πριν από 35 χρόνια, όταν ε, από κοινού ανακτούσαμε την ελευθερία και την αξιοπρέπεια μας στη χώρα μας. Αν σε έλεγε κάποιος ότι σε 35 χρόνια εγώ θα προεδρεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσύ θα είσαι συγκέντρια και θα σου δίνω το λόγο, κανείς δεν θα μας πίστευε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φαίνεται ποια ήταν η πρόοδος αυτή, όχι μόνο της ελευθερίας στη χώρα μας, αλλά της ελευθερίας γενικότερα στην Ευρώπη, μαζί με την Ευρώπη. Έχεις ε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καλημέρα σας. Θα σας παρουσιάσω τη σύνοψη των όσων συζήτησε η ομάδα εργασίας 3 για την προστασία των πολιτών και μια ευρωπαϊκή στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Συμπρόεδρος ήταν ο κύριος Μπουσουτήλ, ε, ευρωβουλευτής και η κυρία ε, Ντάβιτσον, ε, βουλευτής από τη Σουηδία και εγώ ήμουν εισηγήτρια. Στην αρχή της συνεδρίασης τονίσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ακόμα πιο σημαντική η συνθήκη της Λισαβόνας και ο θεμελιώδης χάρτης ε, των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πλέον νέο ρόλο και τα εθνικά κοινοβούλια και περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξ όσων ακούσαμε στη συνεδρίαση αυτή και στην προηγούμενη Ολομέλεια, εκφράστηκαν ουσιαστικά δύο σχολές, ε, σχολές σκέψης και στην ομάδα εργασίας. Περίπου μισή-μισή ήταν ομιλητές. Εντάξει, δεν είναι αριθμητικά αυτά τα στοιχεία. Ορισμένοι λοιπόν επιμένουν πιο πολύ στο να ενισχυθεί ε, η ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, μετά το Μαστρίχ δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι Οι απαιτήσει ασφαλεία δεν ε, μπορούν ποτέ, δεν επιτρέπεται ποτέ να αποδυναμώνουν το σύστημα ελευθεριών και δικαιωμάτων και μάλιστα των ατομικών δικαιωμάτων. Η συζήτηση ήταν πολύ εντατική, πολύ εκτατική και πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, συμμετείχαν πολύ πήραν το λόγο πολλοί οι βουλευτές. Ο κύριος Ποντέχ, ο Γιόνκρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κύριος Κοέγιο Ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της Ρουμανικής Γερουσίας, από το Βελγικό Κοινοβούλιο επίσης συνάδελφοι, την Πολωνική Γερουσία, ο Λόρδος Χάρισον από ε, τη Βουλή των Λόρδων της Μεγάλης Βρετανίας, η κυρία Ζήση από τη Βουλή των Ελλήνων, ε, κάποιος βουλευτής από την Τσεχική Δημοκρατία, από την Αυστρία, τη Φιλανδία, πολλοί συνάδελφοι, πάνω από 20 μίλησαν, εν πάση περιπτώσει. Και ουσιαστικά ε, με κάποιες αποχρώσεις πάντα και ε, όλοι οι ομιλητές επίμειναν σε αυτό ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ε, μεταξύ των ελευθεριών και της ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και εκκρεμούν ήδη από την εποχή του Τάμπερε και της Χάγης. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι πάρα πολύ ευρύ ενδεχομένω και πάρα πολύ ανοιχτό σε κάποια θέματα. Δεν είναι αρκετά περιοριστικό. Καλό θα ήταν στα πλαίσια του προγράμματος ε, χόλμη να αξιολογήσουμε όλε τι πολιτικέ που προέρχονται από προηγούμενα στάδια, γιατί χρειάζονται συγκεκριμενοποίηση και αποκριστάλλωση, αν θέλετε. Επίση θα σα έλεγα ότι από όλε τι παρεμβάσει. μπορούμε να κρατήσουμε ότι η ετοιμιγορία, για να το πω έτσι, για το πρόγραμμα της Στοχόλμης είναι πάρα πολύ θετική. Όπως σας είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει να έχουμε περισσότερη ε, συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ευρύ το πρόγραμμα. Εγώ όμως θεωρώ ότι αν δεν είμαστε φιλόδοξοι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουμε ούτε να φτάσουμε στα επιθυμητά και προτινόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη, τίθεται το θέμα της κατάρτισης της αστυνομίας, της συνεργασίας, των δεδομένων και στοιχείων εγκληματικότητας, πρόσβαση ενώ των διαφόρων ε, αρχών των κρατών μελών, αστυνομικών αρχών και διαφύλαξης της τάξης, συνεργασία μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας των κρατών μελών. Όλα αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Εκπρόσωπος της ε, Βρετανικής Βολής των Λόρδων αναφέρθηκε σε πολύ περίεργες καταστάσεις, έτσι, εξωφρενικές. Γιατί ότι κάνει ερωτήσεις στα αγγλικά, ας πούμε, αστυνομία και περιμένει από τους ε, κακοποιούς, ας πούμε, ή από τους ε, ανθρώπους που έχουν συλλάβει να, να τους καταλάβουν και να τους απαντήσουν στα αγγλικά. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν γίνεται αυτό. Ε, όλα αυτά τα συζητήσαμε, το οργανωμένο έγκλημα, τη συνεργασία στην ανάπτυξη και τη συνεργασία στην ε, ασφάλεια. Ενδιαφέρονται όλα αυτά. Λοιπόν, όλες αυτές τις πολύ σημαντικές προκλήσεις, επαναλαμβάνω, ε, εγγύησεις, δικαιώματα των πολιτών, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης η συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ασφάλεια στην Ευρώπη και να καταπολεμήσουμε τη ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, τις προκαταλήψεις κατά των ομοφιλοφίλων όλα αυτά είναι ε, αξιόπινες ε, πράξεις που στρέφονται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης θέλουμε την Ευρώπη τη συνεργασία στο άσυλο. Κοινή πολιτική μετανάστευση. Πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου. Άλλες προκλήσεις, ε, ε, ε, κρίζωση και πρόληψη νέων και παλαιών αξιόπιων πράξεων που έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Ας πούμε, συνεργασία στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με κάθε μορφή, καταπολέμηση του εμπορίου τρόπου του τράφικινγκ, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, πειρατεία στη θάλασσα, το έγκλημα στο διαδίκτυο, παιδική πορνογραφία και πειρατεία βία κατά των παιδιών, στο σπίτι, στην οικογένεια, στα σχολεία, στις γειτονιές. Αυτά πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ συνοπτικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση και ελπίζω να είναι χρήσιμη για όλους. Και σύντομα να έρθει όχι μόνο το πρόγραμμα της Στοχόλμης, αλλά και η συγκεκριμενοποίησή του στην Ισπανική Προεδρία ενδεχομένω το πρόγραμμα δράση που θα το ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις εισηγητές, παρουσιαστές των αντίστοιχων ομάδων. Οι παρουσιάσεις τους ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και συνεισφέρουν στην συζήτηση την οποία κάνουμε. Τώρα θα περάσουμε στην παρέμβαση της Υπουργού Δικαιοσύνης της Σουηδίας, την κυρία Μπεατρίς Άσκ. Όταν ζητώ από ένα μέλος της σουηδικής κυβέρνησης να πάρει το λόγο, διαπιστώνω ότι η Σουηδία για πάρα πολλά χρόνια και κατά τη διάρκεια πολλών κυβερνήσεων ήταν ένας φάρος ελπίδας για το σύνολο της Ευρώπης, ιδιαίτερα για αυτούς στην Ευρώπη οι οποίοι έπρεπε να μάχονται για την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους. Η χώρα σας ε, έχει ένα παρελθόν που έλεγε πάρα πολλά στους πιο πολλούς από εμάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρτίνες για αυτήν σας την εισαγωγή. Κύριε Μαρτίνες, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε Μπαρό, θα αρχίσω ευχαριστώντας σας για την πρόσκληση στη συνάντηση εδώ με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Χαίρομαι που βλέπω τόσο πολλούς εδώ παρόντες και ιδιαίτερα γιατί μεταξύ των θεμάτων είναι και το πρόγραμμα της Στοκχόρμης. Το πενταετές εκείνο πρόγραμμα που θα συνεχίσει την προσπάθεια της Χάγης. Το όραμα του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής Ευρώπης όπου θα υπάρχει προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων γιατί νομίζουμε ότι το επίπεδο του πολίτη πρέπει να είναι αυτό που καθορίζει όλα τα νομοσχέδια. Η συνεργασία που προβλέπεται πρέπει να είναι κάτι που το γνωρίζει και το ποθεί ο πολίτης, το άτομο. Και γι' αυτό πρέπει να τα νομοσχέδια και τα προγράμματα που εγκρίνονται να έχουν απτές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η καταπολέμηση του εγκλήματος είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό γιατί οι πολίτες ελπίζουν η ευρωπαϊκή συνεργασία να συνεισφέρει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ότι θα αυξηθεί δηλαδή η διάσταση ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της ασφαλείας και της νομικής βεβαιότητας πρέπει να συμβαδίζουν πάντοτε με το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Το διεθνές, η διεθνής εγκληματικότητα είναι κάτι το προφανές ε, ως πρόβλημα, όπως η λαθρεμπορία ναρκωτικών. Σήμερα το πρωί στο BBC στην τηλεόραση ακούστηκε ότι στην, στην Αγγλία υπάρχει εκμετάλλευση παιδιών από εγκληματίες και σεξουαλική τους κατάχρηση. Εκμετάλλευση. Οι πολίτες απαιτούν την καταπολέμηση τέτοιου είδους φαινομένων. Στη Σουηδία ε, εξετάστηκαν όλα αυτά, έγινε μια μελέτη, αλλά υπάρχουν όλο και πιο καινούργιες μορφές εγκληματικότητας, παραδείγματο χάρη μέσω του διαδικτύου. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη δεν ασχολείται καθόλου με θέματα εθνικών συνόρων και γι' αυτό η λύση του προβλήματος αυτού πρέπει να είναι και αυτή διεθνής. Δεν πρέπει τα σύνορα να μας εμποδίζουν να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα. Η συνεργασία λοιπόν σε αυτό το τομέα είναι κάτι το ουσιώδες και προφανές. Πρέπει τα κοινοβούλια να ελέγχουν βέβαια εάν πράγματι υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία. Αυτό είναι βασικά το πρόγραμμα της Στοχόλμης, να βρεθούν κοινέ λύσεις για κοινά προβλήματα μεταξύ των οποίων και πιο αποτελεσματικά συστήματα για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών και σίγουρες μέθοδοι για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι πληροφορίες για το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να γίνονται γνωστές, να διαδίδονται. Την 1η Οκτωβρίου η Σουηδική Προεδρία σε συνεργασία με την Europol οργάνωσε μία υπουργική συνάντηση στη Χάγη για αυτού του είδους την αστυνομική συνεργασία γιατί ο στόχο τη Europol, ο σκοπό της Europol είναι ακριβώ να διευκολύνει τη μαθεωριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματο. Είπα και πριν ότι σημαντικό τμήμα της διαμεθοριακής συνεργασίας είναι και η ανταλλαγή πληροφοριών που διαθέτουμε για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά σε πανενωσιακό επίπεδο θα έπρεπε να στοχεύσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών για να είναι αποτελεσματικότερη. Επίσης φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υπάρχουν εγγυημένα ελάχιστα πρότυπα για, κατά την ανταλλαγή αυτή για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες αλλά δεν είναι συνδυασμένες δεν έχει νόημα. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια ασφαλής Ευρώπη με αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος αλλά και σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι κάτι το δυνατόν <clears throat> και πρέπει να συνδυαστούν τα δύο ταυτόχρονα να ε, υπάρχει σεβασμός και των δύο αρχών. Η αμοιβαία αναγνώριση είναι επίσης ε, μια σημαντική πτυχή. Για να υπάρχει κάτι τέτοιο αποτελεσματικά πρέπει η συνεργασία Πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων δικαστικών συστημάτων. Αλλά είναι και θέμα του αισθήματο που πρέπει να έχουν οι πολίτες ικανοποίησης για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών αυτών. Παραδείγματο χάρη, η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων είναι κάτι το ουσιώδε. Έτσι αυξάνεται όντω η εμπιστοσύνη. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη και περισσότερη γνώση, πληροφόρηση για τα δικαστικά συστήματα μεταξύ των χωρών μέσω του Εράσμου ή δικτύων που υπάρχουν ήδη και των μηχανισμών αποτίμηση, εκτίμηση αμοιβαίας αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. Ίσως το κυριότερο μέσο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι να υπάρξουν περισσότερες εγγυήσεις ως προς την ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη του καθενός. Απλά πράγματα όπως την χορήγηση της πληροφόρησης προς κάποιον κατηγορούμενο στη γλώσσα την οποία καταλαβαίνει και των θυμάτων, όχι μόνο των κατηγορουμένων. Με χαρά διαπίστωσα ότι το Συμβούλιο δέχτηκε ένα πρόγραμμα για τα δικαιώματα αυτά των κατηγορουμένων και των θυμάτων. Από το 2007 είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις αλλά φαινόταν ότι δεν θα ήταν πιθανή η συμφωνία και όμως υπήρξε. Κάθε πρόγραμμα που είναι σωστά στοχευμένο και προσέχει την προστιθέμενη αξία που πρέπει να βλέπει ο πολίτης στην καθημερινή του ζωή θα πετύχει. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα την άποψη των θυμάτων. Η αυξανόμενη κίνηση των πολιτών από χώρα σε χώρα σημαίνει ότι πρέπει να μπορούν οι πολίτες να έχουν πληροφόρηση σε γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν αν έχουν κατηγορηθεί ή αν έχουν υποστεί κάποιο έγκλημα. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη, τη δικαστική διαδικασία. Και οι αποζημιώσεις που θα αποφασίζονται να είναι ανάλογες με το έγκλημα. Δικαιώματα λοιπόν των θυμάτων εγκλημάτων. Η βοήθεια στα θύματα πρέπει να αυξηθεί και το πρόσεχε αυτό ιδιαίτερα το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Τον προηγούμενο μήνα η Προεδρία υπέβαλε την πρώτη μορφή του εγγράφου, του σχετικού εγγράφου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας και η σχετική δήλωση της Επιτροπής κάνει μία σύνοψη των πρώτων του συμπερασμάτων. Προσθέσαμε από τότε ένα κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις γιατί πολλές χώρες μέλη μας το επέστησαν αυτό ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις διαπραγματεύσεις μας πρέπει πράγματι να το σκεφτούμε περισσότερο. Η σύνδεση μεταξύ των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικών είναι κάτι που πρέπει επίσης να ενισχυθεί γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξωτερική διάσταση δεν πρέπει να ξεχαστεί στο Κορεπέρ κάθε εβδομάδα το συζητούμε και στις 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου στην Υπουργική Διάσκεψη θα ξανασυζητηθεί το θέμα το οποίο τελικά θα συζητηθεί και από το Κοινοβούλιο, ε, του προηγουμένως μάλλον στις 26 Νοεμβρίου. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει αλλαγές για θέματα ατομικών δικαιωμάτων, νέα νομικά υπόβαθρα για ορισμένες διαδικασίες προβλέπεται αυξημένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι και τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν νέα καθήκοντα από τη συνθήκη της Λισαβόνας διότι οι πολίτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ. Και τώρα θα μιλήσει ο Επίτροπος, ο φίλος μας κύριος Παρό, για δέκα λεπτά. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μπεατρί Σάσκ, η Προεδρεύουσα, του Συμβουλίου σας εξέθεσε τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος της Σουηδικής Προεδρίας. Εκ των προτέρων θα ήθελα να υπογραμμίσω και το κάνω αυτό την παρουσία του Περ Βέστερμπεργκ, τον ρόλο τον οποίο παίζει η Σουηδική Προεδρία, ένα πολύ θετικό ρόλο, ο οποίος μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε ένα πρόγραμμα στο Κόλμιτς ιδιαίτερα φιλόδοξο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Λόπε Αγουιλάρ και τους δύο άλλους ε, συνεισηγητές του για τα στοιχεία που μας έδωσαν. Θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του προγράμματος της Στοκόλμης σε μια φάση όπου θα κληθούμε να εφαρμόσουμε τα στοιχεία τα οποία προβλέπει για τον τομέα μας η συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιτρέψουν ο τομέας που μας ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο και να δραστηριοποιηθεί και το ίδιο το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο όταν συμμετέχει στις διαδικασίες ως συνομοθέτης προσφέρει θα έλεγα υψηλή προστιθέμενη αξία. Έχω εμπειρία αυτού που λέω και σαν επίτροπος για τις μεταφορές και το βιώνω και σήμερα στα πλαίσια των μεταναστευτικών πολιτικών ή των συζητήσεων με το Κοινοβούλιο για τις μεταναστευτικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν εκφράζω την χαρά μου γιατί βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντάσσεται πλήρως στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής της κοινότητας δικαίου την οποία όλοι επιθυμούμε. η διεύρυνση της χρήσης της <clears throat> ειδική πλειοψηφίας στο Συμβούλιο θα μας επιτρέψει ελπίζω να ξεπεράσουμε κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Συν τη άλλη, η συνθήκη τη Λισαβόνα βελτιώνει και την θέση των κοινοβουλίων των κρατών μελών στα πλαίσια τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτό θα μα επιτρέψει να κάνουμε ακόμα πιο σεβαστή την αρχή τη επικουρικότητας, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σε θέματα πάρα πολύ σημαντικά όπως το ποινικό και το οικογενειακό δίκαιο είναι σαφές ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να αγνοηθεί όπως δεν μπορεί να αγνοηθούν και οι διαφορετικές βέβαια νομικές παραδόσεις. Ευχαριστώ πάντως τους συναδέλφους από τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών για την συνεισφορά τους στην κοινή προσπάθεια. Είναι αλήθεια ότι στα πλαίσια της κατάργησης και του τρίτου πυλώνα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να προσφύγουμε στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα βήματα προόδου του κράτους δικαίου ή μάλλον της Ευρώπης του δικαίου θα γίνουν πραγματικότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης, στα πλαίσια της προσπάθειας εφαρμογής του προγράμματος της Στοχόλμης, θα προχωρήσουμε και στην επόμενη, θα έλεγα, θεσμική βάση, η οποία θα οδηγήσει ακριβώς σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της κοινότητας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία από την οποία προσδοκά τόσα ο Ευρωπαίος πολίτης. Αγαπητή κυρία Άσκ, εμείς θέσαμε τον πολίτη στο κέντρο αυτού του προγράμματος. Το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι φιλόδοξο, αλλά είναι και ιδιαίτερα συνεκτικό και είναι αντικείμενο θα έλεγα πνεύματος συνεργασίας. Χαρακτηρίζεται μάλλον από το πνεύμα συνεργασίας όλων και έχω την εντύπωση ότι και η ανακοίνωση της Προεδρίας θα είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες οι διαπραγματεύσεις και σε επίπεδο κορεπέρ, όπως είπε η κυρία Άσκ. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις καθόλου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι το Συμβούλιο ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στα μέσα Δεκεμβρίου. 11 και 12 Δεκεμβρίου θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις. Θα ήθελα τώρα πάρα πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια από τα στοιχεία της πολιτικής που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ε, να προωθήσουμε και θα επαναλάβω ίσως κάποια από αυτά τα οποία ε, είπε η κυρία Άσκ. Καταρχάς, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι προφανές ότι η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν αναιρεί τίποτα και δεν αφαιρεί τίποτα από την εθνική θα έλεγα αντίστοιχη. Προσθέτει κάποιες νέες διαστάσεις όπως την ελευθερία διακίνησης στην οποία νομίζω θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι μια πραγματικά σημαντική μορφή ελευθερίας Έχουμε τη διασφάλιση επίσης και της ιδιωτικής ζωής μέσω της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και εδώ η Ευρώπη θα πρέπει να έχει στη διάθεσή, σας, στη διάθεσή της μια ουσιαστική αρχιτεκτονική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προϋποθέτει αυτή η ευρωπαϊκή αν θέλετε ε, ιδιότητα του πολίτη και μια δυνατότητα συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη καλύτερη από ό,τι σήμερα και ίσως και την καθιέρωση ε, μία συγκεκριμένη ημέρα για όλους που θα μπορούσε να είναι η 9η Μαΐου για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο πρόεδρος Λόπες Αγκουιλάρ, εμπλουτίζεται αυτή η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη από διαφορετικά χαρακτηριστικά και έχουμε επίσης και την ε, δυνατότητα πλέον σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσουμε και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Για τη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ που εμένετε στην κατάργηση του εξεκουάτορ. Εάν πράγματι θέλουμε να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη, θα πρέπει να απομακρύνουμε τα εμπόδια τα οποία έχουμε μπροστά μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του επιμένει ιδιαίτερα στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Η αρχή βέβαια της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να είναι ο ακαγωνιαίος λίθος της δημιουργίας αυτής της Ευρώπης της δικαιοσύνης. Και αυτή η αμοιβαία αναγνώριση, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη όλων των συμμετεχόντων ε, στα εκτενόμενα της δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει κοινοί κανόνες, και θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να είναι σε θέση σύντομα να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που τους παρέχει η δικαιοσύνη σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει άλλωστε και η ενίσχυση αυτή της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης ή της ευρωπαϊκής διάστασης της δικαιοσύνης να στηρίξει και την σωστή λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας. Τρίτος άξονας η ασφάλεια. Έχουμε ανάγκη από μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να παραμένει συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα θεμελιώδη συγγνώμη δικαιώματα. Είναι μια σφαιρική θα έλεγα, έχει σφαιρικές ιδιότητες αυτή η στρατηγική. Εδράζεται στην αστυνομική συνεργασία, στην συνεργασία σε επίπεδο ποινικού δικαίου ή ποινικής δικαιοσύνης αν θέλετε και τέλος σε μια σωστή διαχείριση της πρόσβασης στο ευρωπαϊκό έδαφος, έλεγχο συνόρων δηλαδή. Και τέλος, τέταρτο κεφάλαιο, είναι το θέμα της μετανάστευσης. Η μετανάστευση απαιτεί και την αλληλεγγύη με, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τη συνεργασία, μια εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες. Αυτές οι δύο πολιτικές θα πρέπει να εγγραφούν σε ένα πεδίο μακροπρόθεσμο προϋποθέτουν από τη μία την ενασχόλησή μας με σωστό τρόπο με την νόμιμη μετανάστευση που παρέχει στους ε, τακτικούς ή τακτούς μετανάστες αν θέλετε ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες και ταυτόχρονα ένα όχι στην παράνομη μετανάστευση και σε όλες τις εγκληματικές παράπλευρες δραστηριότητες. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την Ευρώπη του ασύλου, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάθε προσώπου που ζητά πολιτικό άσυλο, ζητά την προστασία και πρέπει να παρέχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας όταν τα χορηγούμε. Αυτά είναι λοιπόν τα τέσσερα βασικά κεφάλαια τα οποία θα επιτρέψουν η Ευρώπη μας να προχωρήσει σαν κοινότητα δικαίου στην υπηρεσία του πολίτη. Θα υπάρξει λοιπόν το πρόγραμμα της Στοχόλμης, υπάρχει και το πρόγραμμα δράσης στο οποίο θα υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι πλέον ο ρόλος των κοινοβουλίων, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθεί και θα σας επιτρέψει σε εσά όλους τους βουλευτές και ευρωβουλευτές να μπορέσετε να συνεισφέρετε σε αυτή την τεράστια προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός μιας κοινότητας δικαίου και νιώθω μέσα από την προσπάθεια που γίνεται και αυτές τις δύο μέρες την προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει για τη δημιουργία μιας Ευρώπης δικαίου, μιας Ευρώπης του πολίτη. Αυτά πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για αυτά τα λίγα λόγια. Και τώρα Απευθύνομαι και στη συνάδελφο την κυρία Υπουργό και θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας και ίσως απαντήσουμε και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρό. Όπως πάντα αξίζει να υπογράψουμε, να υπογραμμίσουμε συγγνώμη. Ότι όλα αυτά τα χρόνια έχετε δείξει ότι είστε μέγας φίλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατανοείτε πάρα πολύ ε, τα μελήματά μας και είναι πολύ καλή ευκαιρία να σας αποτίσουμε ένα φόρο τιμής γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα θα παραδώσω την Προεδρία στον συνάδελφο Βέστεμπερκ. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση η δυνατότητα που μου δόθηκε να προεδρεύσω εδώ στη διάσκεψη με όλους σας. Κύριε Βέστεμπερκ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι μόνο με το σχετικό έντυπο μετά την υποβολή του σχετικού γράφου θα χορηγείται ο λόγος. Όποιος θέλει να θέσει ερώτημα πρέπει να λέει και σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα, στην Υπουργό ή σε κάποιον άλλον ή στον Επίτροπο Μπαρό. Και στο τέλος θα δοθούν απαντήσεις. Επίσης ο χρόνος ομιλίας είναι μόνο τρίλεπτος Αρχίζει λοιπόν ο γύρος. Η κυρία Ντέιβιντ από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Δεχόμαστε μεν το στόχο του προγράμματος της Στοκόλμης για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης ασφαλείας και ελευθερίας και δικαιοσύνης αλλά οι πτυχές ασφαλείας του προγράμματος αυτού μας ανησυχούν γιατί μπορεί να καταλήξουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης φρουρίου. Παρά το ότι μας καθησυχάζουν για την ανεξαρτησία με την οποία θα γίνει ο έλεγχος των φακέλων και των στοιχείων των προσωπικών, πρέπει ακόμη να βρεθεί τρόπο συνδυασμού της ασφάλειας με το σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο συνδυασμός των στοιχείων από τις διάφορες χώρες πρέπει να γίνει με πλήρη ορατότητα και διαφάνεια η Ευρώπη δίνει όντως την εντύπωση ότι απλώς προστατεύει τον εαυτό της και δεν εφαρμόζει τις αρχές αλληλεγγύης και ελευθερίας ή δικαιοσύνη που υπενθυμίσαμε χθες στο εργαστήριο υπαριθμών 1. Οι ομάδες ταχείας παρέμβασης και η γαλάζια κάρτα αποκλείουν από πολλούς αποκλείουν πολλούς που θέλουν να φύγουν, να ξεφύγουν από τις συνθήκες όπου ζουν και αυτοί στο εξής θα κρίνονται σε φυλακές και κέντρα κράτησης. Γι' αυτό οι κομμουνιστές βουλευτές καταδικάζουν την επιλεκτική και καταπιεστική αυτή πολιτική μετανάστευσης. Ο εισηγητής Λοπές Αγγιλάρη είχε πει χθες στα συμπεράσματά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μία νέα κοινή βάση, ένα νέο κοινό παρονομαστή, αλλά δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε δικαιώματα ούτε ταυτότητες. Το θύμισε και ο κύριος Μαρό προηγουμένως. Με αυτό συμφωνούμε, γιατί για μας η ποικιλομορφία που δημιουργεί η μετανάστευση είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό, είναι ένας πλούτος που διαθέτουμε και πρέπει λοιπόν να δώσουμε στους μετανάστες αυτούς δικαιώματα, όποια και να είναι η προέλευσή τους. Καταλήγω λέγοντας ότι παραμένουν ανησυχίες για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ο στόχος οικοδόμησης μιας Ευρώπης ασφαλείας δικαιοσύνης και ελευθερίας μπορεί τελικά να μας απομακρύνει από την Ευρώπη που θέλουμε ισότητας δικαιοσύνης και αδελφοσύνης μιας Ευρώπης, από μια Ευρώπη των λαών δηλαδή που θα έπρεπε να εγγραφεί και αυτή στο πρόγραμμα της Στοκόλμης. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο Αλμπέρτος Μαριτάτε από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. παρακολούθησα και τις εργασίες της ομάδας ε, εργασίας στην οποία συμμετείχα και διαπίστωσα ότι τα σχόλια τα οποία έγιναν ήταν μεταξύ τους αρκετά συνεκτικά και νομίζω ότι και οι επόμενες συναντήσεις θα πρέπει να είναι ε, πιο συγκεντρωμένες σε ένα-δύο θέματα και πάνω σε αυτά τα θέματα να προσπαθήσουμε να ε, συνεισφέρουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο κοινοβούλια μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, να αναφερθώ σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα, το μεταναστευτικό. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαχειριστεί και να ελέγξει το μεταναστευτικό φαινόμενο. Δεν μπορεί η πολιτισμένη Ευρώπη να δείχνει τους μύστης και να απειλεί με τη δύναμή της αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν από το θάνατο και από τον κίνδυνο γενικότερα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με γενικό τρόπο. Θα πρέπει να ελέγξουμε το φαινόμενο αυτό να συνδυάσουμε την καταστολή με την πρόληψη, να κάνουμε συγκεκριμένες συμφωνίες σωστά στοχευμένες ε, με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτές οι μεταναστευτικές ροές, να προετοιμάσουμε σε επαγγελματικό επίπεδο και σε πολιτιστικό επίπεδο όλους αυτούς οι οποίοι σκοπεύουν να έρθουν στην Ευρώπη έτσι ώστε να καταφέρουμε να μετριάσουμε σε επίπεδο πολιτισμικό τις συγκρούσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς και ταυτόχρονα να ασχοληθούμε με αυτήν την πολύ ευαίσθητη στιγμή σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θα να σεβαστούμε, να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με αυτά τα κέντρα παραμονής που άλλαξαν όνομα μένα αλλά δεν πάβουν να παραμένουν και να είναι διοικητικά κρατητήρια ή φυλακές. Αυτοί οι χώροι θα πρέπει να είναι όχι κέντρα διερχομένων για αυτούς οι οποίοι θα επαναπροωθηθούν στις χώρες τους, αλλά πραγματικά κέντρα υποδοχής ή έστω και κέντρα προετοιμασίας για αυτούς στους οποίους θα υπάρξει, θα δοθεί μια κάποια συνδρομή για να επιστρέψουν με τη δική τους θέληση στις χώρες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και εμείς στη χώρα μας, η οποία προσπαθεί κυρίως να αντιδράσει σε κατασταλτικό επίπεδο Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια ε, γιατί όπως ξέρετε θεωρείται έγκλημα η μετανάστευση η παράνομη. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν χρησιμεύει για να μετριαστεί το συγκεκριμένο μεταναστευτικό φαινόμενο, απλά παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. δικαιώματα συγγνώμη. Η συνδρομή στην επιστροφή, οι συμφωνίες υποστήριξης και βοήθειας προς τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, Αυτό είναι ο ρόλος τον οποίο πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη, μια Ευρώπη πολιτισμένη που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουσουτήλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς, όπως και ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες, να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τον Επίτροπο Μπαρό για όσα έχει κάνει στον τομέα αυτόν και γιατί τόλμησε να προσδιορίσει τι ακριβώς χρειάζεται ακόμη να γίνει για να επιτευχθεί ο χώρος ελευθερίας και δικαιοσύνης. Εγώ την εσωτερική αγορά τη θεωρώ ως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τα επόμενα χρόνια ίσως η δημιουργία αυτού του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας να είναι η επόμενη μεγαλύτερη πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη καταλαβαίνουμε αμέσως πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Από τη θετική πλευρά, η συνθήκη της Λισαβόνας που σε λίγο θα τεθεί ενισχύει θα μας δώσει τα εργαλεία που να μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε το στόχο αυτό. Γιατί η λήψη των αποφάσεων με πλειοψηφικό τρόπο θα, ε- υποχρεώσει, θα μας υποχρεώσει όλους να είμαστε πιο επικοδομητικοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η συνθήκη λοιπόν της Λισαβόνας θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, πιο απτά, τη δημιουργία αυτού του χώρου ελευθερίας κλπ. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες και ευαισθησίες ανάλογα με τις ομάδες και όχι μόνο τις ομάδες, αλλά και μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών της Ένωσης. Και αυτό δεν σημαίνει ότι καταλήγουμε σε παράλυση, αλλά ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την επίτευξη συμβιβασμών. Όσοι ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μερικοί ενδιαφέρονται κυρίως για την τρομοκρατία, άλλοι για τις πολιτικές ελευθερίες, άλλοι για την παράνομη μετανάστευση και άλλοι για τα δικαιώματα των μεταναστών. Πώς θα βρούμε την ισορροπία λοιπόν. Πριν από μερικές μέρες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε σε μια πολύ αμφιλεγόμενη απόφαση για την επίδειξη του εσταυρωμένου στα Ιταλικά σχολεία. είναι όντως αμφιλεγόμενες οι μέθοδοι και τα θέματα αυτά και δεν είναι εύκολο να συνδυάσει κανείς τις διαφορετικές απόψεις. Είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ή όχι. Χρειάζεται μεγάλο θάρρος. Και στο εξή, τι πρόκειται να γίνει. Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν οι ακροάσεις των μελλοντικών επιτρόπων και θέλουμε να δούμε οι νέες ευθύνες που μέχρι τώρα βάριναν μόνο έναν άνθρωπο τώρα θα βαρύνουν δύο. Ο κύριος Μπαρόσο είπε ότι θα υπάρξει ένας επίτροπος για δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα και άλλος για εσωτερικές υποθέσεις και μετανάστευση. Θέλουμε λοιπόν, προσβλέπουμε στις ακροάσεις για να δούμε τι, διασφα... τι εγγυήσεις θα μας δώσουν οι μελλοντικοί επίτροποι για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να πετύχουν το συνδυασμό των δύο. Έπειτα υπάρχει το θέμα της έγκρισης του προγράμματος της Στοκχόλμης και του σχετικού του συνοδευόμενου προγράμματος δράσης. Η εφαρμογή, ο τρόπος εφαρμογής είναι εδώ το κλειδί. Για πολύ καιρό ακούγαμε λόγια και βλέπαμε έγγραφα, αλλά τώρα αυτό που θα προσέξουμε θα είναι η εφαρμογή. Αν θέλουμε πράγματι να υπάρξει ένας χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας, τότε η εφαρμογή είναι το κλειδί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Θωμάς Γκρούλιτς από την Τσεχική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι παρόντες συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, ανέφερε και ο Επίτροπος, είναι πολύ σημαντικά για μας και θέλω λίγο να τα σχολιάσω. Η Τσεχική Γερουσία έχει λάβει απόφαση αρχής για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ομιλεί για στόχους ρεαλιστικούς. Θα πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά ε, τι πρωτοβουλίες ε, αναλαμβάνουμε και αν έχουν πραγματικά υπεραξία, μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ακούμε συνέχεια ότι το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο. Εντάξει, καλή φιλοδοξία, αλλά θα πρέπει να είναι και εφαρμόσιμο εκτός από φιλόδοξο. Ε, κατά την άποψή μας λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές και οι δικές μας παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης όπως το παρουσίασε η Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο προϋποθέσεις που θεωρεί ε, εκ των όνων κάνευ η γερουσία της τσεχικής δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι επιθυμητό, για παράδειγμα, η Frontex να γίνει ένα είδος ε, στρατού για την εξωτερική φύλαξη των συνόρων, τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων Αυτό που έχουμε σήμερα, ο συντονισμός και η συνεργασία μας αρκεί προς το παρόν. Προστασία των συνόρων θα πρέπει να είναι και να παραμένει ε, αντικείμενο και υποχρέωση των κρατών μελών. Στη συνέχεια, η Τσεχική Δημοκρατία επίσης η Γερουσία ασχολήθηκε με τη μετανάστευση. Η λάθρο μετανάστευση καταπολεμείται προληπτικά. Ενώ στην νόμιμη μετανάστευση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προσαρμογή ε, στις ε, διάφορες ε, αγορές εργασίας στην κάθε χώρα μέλος. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση ό,τι αφορά τα επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές προς τους μετανάστες. Το κείμενο λέγει και προβλέπει ότι οι νόμιμοι μετανάστες θα πρέπει να απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όχι. Έχουμε εδώ κατάχρηση των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και αυξάνεται η μετανάστευση για να παίρνουν τα επιδόματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Μπενιστή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γαλλική αντιπροσωπεία χαίρεται ιδιαίτερα για την κοινή πρωτοβουλία του Σουηδικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής περί της κοινοβουλευτικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφαλείας, Δικαιοσύνης και Ελευθερίας. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και η γαλλική αντιπροσωπεία δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον Επίτροπο Μπαρόν, τονίζει ιδιαίτερα τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ευρωπαϊκού τιούτου, το οποίο θα έχει αυξημένες δικαιοδοσίες μετά τη θέση ενισχύει της συνθήκης της Λισαβόνης. Ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης του οργανωμένου κλίματος σήμερα είναι η προστασία του Ευρωπαίου πολίτη η βελτίωση της συνεργασίας και του αστυνομικού και δικαστικού συντονισμού μέσα στο χώρο του Σέγγεν. Οι επιθέσεις της 11 η Σεπτεμβρίου μας όθησαν να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πρέπει όμως να υπάρξει βελτίωση της διάδοσης αυτής των πληροφοριών της ανταλλαγής που υπάρχουν στα διάφορα αστυνομικά αρχεία είναι ουσιώδες στοιχείο αυτό της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Ε, κανείς δεν θα καταλάβαινε η συνεργασία μεταξύ Ένωσης και, Ευρω... και Ηνωμένων Πολιτειών να υπάρχει ενώ δεν υπάρχει τίποτε αντίστοιχο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Οι τράπεζες δεδομένων έχουν αυξηθεί πολύ από τις αστυνομίες και είναι σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης του εγκλήματος που είναι όλο και περισσότερο οργανωμένο και διεθνές. Πρέπει λοιπόν τα κράτη να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και κυρίως να έχουν αυτόματη και αμοιβαία πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων είτε πρόκειται για στοιχεία του βιολογικά είτε άλλα. Πέρα δηλαδή και από την απόφαση πλαίσιο του 2008. Είναι απαραίτητη η ανταλλαγή αυτή των πληροφοριών και για τα γενετικά στοιχεία. Κύριε Επίτροπε λοιπόν, ερωτώ, προβλέπονται προβλέπεται η χορήγηση των πραγματικών εργαλείων που χρειάζεται η διεθνής αστυνομική και δικαστική συνεργασία για την προστασία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Άντριου Μπρόνς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. μπρονς απο το ευρωπαικο κοινοβουλιο ο Ραμόν Χαουρέγγι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τη Σουηδική ε, Προεδρία. Είναι καταπληκτική ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε αυτό το ζωτικό χώρο ασφάλειας και ελευθερίας για την Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να πω στους συναδέλφους και να θυμίσω ότι ο δρόμος για να προχωρήσουμε προς αυτό το πεδίο είναι γεμάτο ε, αποτυχίες. Θα πρέπει να το θυμηθούμε. Θέλω να σας θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι πριν από χρόνια ήδη όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλησε να ε, ε, ε κάνει μια απόφαση πλαίσιο για να ενοποιήσει λίγο το σύστημα της ποινική δικαιοσύνης μετά από τρία χρόνια εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Οπότε ο δρόμος προς το στόχο αυτό είναι γεμάτος εμπόδια. Για το λόγο λοιπόν αυτό, έχουμε συγκεντρωθεί τώρα όλοι εδώ και το συζητάμε και θα είμαστε πρωταγωνιστές της διαδικασίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω έτσι εδώ όπως έχουμε συγκεντρωθεί τα εξή τέσσερα που μου φαίνονται σημαντικά ως για να τα ακολουθήσουμε. Πρώτον, είναι θεμελιώδους σημασίας το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσουν στεναρή την αρχή της πρωτοβουλία. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία, ουσιαστικά δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Συνιστώ λοιπόν και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρουν στο Κοινοβούλιο προτάσεις. Να μας κάνουν προτάσεις για κανόνες που σιγά σιγά να συμπλησιάζουν τα ε, ε, συστήματα ποινική δικαιοσύνη και ποινική δικονομίας. Θέλω να πω και στην κυρία Άσκα επίση, δεύτερο, ότι χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη, γιατί είναι μεγάλη τεχνική περιπλοκότητα αυτών των νομικών κανόνων και θα μα οδηγήσουν στην ανάγκη να αναγνωρίσουμε ένα στα συστήματα του άλλου τη δικαιοσύνη ποινική δικονομίας, αστυνομία, εργαστήρια, συστήματα επιστημονική ε, ανείχνευση, ε, αποτυπωμάτων, σήμανση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να συμμετέχουν πραγματικά και να συνεργάζονται οι χώρες. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη, α πούμε, οι Γερμανοί στου Έλληνε. Ε, ή το ιατροδικαστικό εργαστήριο της Λιθουανίας δεν εμπιστεύεται το ισπανικό σύστημα, το δικαστικό, δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η αρχή της αμοιβέ εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, αρχή της ισορροπίας. Η ισορροπία, λέγω, μεταξύ της παλιάς αυτής διαμάχης ε, ασφάλειας και ελευθερίας και η διελκυστίδα αυτή. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν είναι ότι φέρει την αρχή της ασφάλειας και το κοινοβούλιο την αυθεντία της ελευθερίας. Όχι. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις προτάσεις που κάνει η εκτελεστική εξουσία και τα κοινοβούλια. Εμείς οι βουλευτές δεν είμαστε οι μόνοι θεματοφύλακε τη αρχή των συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα τέταρτο Κάτι που είπα και χθε να υπενθυμίσω. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε εάν δεν υπάρχει η αρχή της εκχώρησης, της γενεοδορία, της μεγαλοψυχίας. Αν λέει ε, το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο κάτω τα χέρια αυτό είναι δική μου αποκλειστική αρμοδιότητα, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ. Δεν θα μπορέσει ποτέ να οικοδομηθεί αυτή η πολιτική βούληση που έχτισε την Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Η Ευρώπη έχει γίνει με εκχωρήσει, με γενεοδορία, με παραχωρήσει, με αναγνώριση ότι θα πρέπει να χτίσουμε την Ευρώπη, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που νομοθετεί για όλους. Αυτό ο άξονας λοιπόν της ασφάλειας και της ελευθερίας έχει μεγάλη δυσκολία, περιπλοκή, δικονομική, ποινική, δικαστική και το έχουμε αυτό το έργο μπροστά μα. Γι' αυτό ε, απαιτεί και καλεί σε αυτή την αρχή της γενεοδορίας για εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Μια πολιτική βούληση για να αναπτυχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Ιγνάσιο Κωσίδα Γουτιέρες από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Επίτροπο Μπαρό και την Υπουργό κυρία Άσκ για την όθηση που δίνουν σε αυτή την υπόθεση της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης με το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Ωστόσο, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω για τρεις κινδύνους που ενδεχομένως να βρούμε μπροστά μας στην οικοδόμηση Πρώτος κίνδυνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερες εξουσίες ε, από αυτό που του επιτρέπουν οι ίδιες τις ιδιαιτότητες, Δηλαδή να, να δημιουργήσει προσδοκίε ότι θα αναλάβει μεγάλες ευθύνες και θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών. Ενώ είναι σημαντική αρχή ότι η ευθύνη αυτή είναι των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίζει ένα χώρο, θα βάζει κοινού κανόνε. Ε, θα πρέπει να ενισχύει τη συνεργασία και να δημιουργεί τα όργανα και τα μέσα γι' αυτό. Αλλά οι πρωταγωνιστές και αυτοί που παίζουν στο παιχνίδι τη ασφάλεια, παραμένουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερη προειδοποίηση. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την περισσότερη ασφάλεια με περισσότερη γραφειοκρατία. Καμιά φορά έχει διδάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε έχει πρόβλημα να δημιουργεί ένα οργανισμό και το πρόβλημα επιπλέκεται την αλληλένεται. Δηλαδή, να μην ζητήσουμε τώρα, δεν στηρίζουμε την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής αστυνομίας. Αυτό που χρειάζεται είναι αποτελεσματικά εργαλεία για να συνεργάζονται μεταξύ τους οι αστυνομίες. Και τελευταία προειδοποίηση για τον τρίτο κίνδυνο. Επίσης, κινδυνεύουμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα οχυρό, μπούνκερ δηλαδή. Γιατί είναι χήμερα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε μια Ευρώπη πιο ασφαλή σε έναν κόσμο που είναι όλο και πιο ανασφαλής. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να ρίξουμε τα εμπόδια που ε, κάνουν την εσωτερική, ένωση, την εσωτερική ασφάλεια να αποτελματώνεται. Όταν μιλάμε για ε, την απειλή από την τρομοκρατία αυτή αφορά και τις πόλεις μας και το Αφγανιστάν ή όταν μιλάμε για την καταπολέμηση των ναρκωτικών ε, δεν είναι μόνο τα καρτέλ της Κολομβίας αλλά και στην Αφρική ε, είναι το πρόβλημα. Ε, από διάφορα αποτυχημένα και χρεοκοπημένα κράτη. Έτσι, θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και τις μεγάλες προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάση από το Φινλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σουηδία, γιατί είναι καταπληκτικό για μένα το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Και καλή συνέχεια του προγράμματος του Τάμπερε και της Χάγης. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, πιστεύω, χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαπιστώνουμε ότι στο χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας στην Ευρώπη έχουμε στόχους φιλόδοξους. Πρέπει να βελτιώσουμε όμως πολύ ε, τη δράση μας. Αν συγκρίνουμε τι κάνουμε εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε φοιτητή γνωρίζει απ' έξω το Σύνταγμα και ξέρει τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο. Επιπλέον το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις που έχουν και φιλοσοφική αιτιολόγηση και ε, εξήγηση κάθε φορά. Στην Ευρώπη όμως πολλές φορές έχουμε προβλήματα με την επιχειρηματολογία και την αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων. Εγώ θυμάμαι ότι στη Σοβιετική Ένωση γινόταν λόγος για διάφορες δημοκρατίες. Σοβιετική δημοκρατία, διεθνή δημοκρατία. Προσοχή έτσι με αυτές τις αποχρώσεις των ιδεών και των ενιών γιατί μπορεί να έχουμε και στρεβλώσεις αλλά και χειραγώγηση. Πρέπει επίση να σα πω ότι πολλέ χώρε διαθέτουν συνταγματικά δικαστήρια που παίρνουν αποφάσει. Έχουμε α πούμε, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο που έχει εκδώσει κάποιε αποφάσει. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσουμε τι αποφάσει αυτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τι μεταφράσουμε στα αγγλικά για να έχουμε σιγά σιγά μια ευρωπαϊκή νομολογία στον τομέα αυτό. Επίση, θα πρέπει να μελετήσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικές αποφάσεις και μας αφορούν όλους. Και στις χώρες μας και στα δικαστήριά μας θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτά τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πώς ε, στοιχειοθετεί τις αποφάσεις του. Όλα αυτά είναι σημαντικά και παραβάνω οι δικαστικές αποφάσεις να έχουν καλή επιχειρηματολογία και αιτιολόγηση για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπίστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως πρέπει. Προσοχή επίσης με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποια διεθνή πρωτόκολλα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάντα θα πρέπει να προσέχουμε και ε, να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το παρατηρητήριο της Βιέννης να έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Τελειώνω, Πρόεδρε. Η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει ε, στην άσκηση της και την επιβολή της δικαιοσύνης. Και τα έγγραφα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι διαφανή και στη διάθεση όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόνς πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά για την Ευρώπη των πολιτών. Συμφωνώ με αυτό. Πράγματι θα ήθελα εγώ να δω μια Ευρώπη ελευθέρων πολιτών και ελευθέρων κρατών. Όχι μια Ευρώπη ε, πολιτών ενός ομοσπονδιακού κράτους, ενός ομοσπονδιακού υπερκράτους. Θα ήθελα επίσης ε, να δω να γίνονται δημοψήφισματα για να αποφασιστεί το αν θα υπάρξει ή όχι αυτό το υπερκράτος. Ακούγονται λόγια πολλά για τη δημοκρατία, πολλά ακούμε για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αλλά τίποτα δεν κάνουμε. Στην χώρα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, στο Βέλγιο, εδώ και λίγα χρόνια, το κράτος πήρε μέτρα για να απαγορεύσει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα. Στην Ουγγαρία ε, εκπρόσωποι των κατασταλτικών δυνάμεων επετέθησαν σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, ε, τους χτύπησαν, τους συνέλαβαν και τους φυλάκισαν. Δεν υπάρχει προστασία ε, της, του ελεύθερου λόγου γενικότερα στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και δεν σεβόμεθα στην Ευρώπη τον ερετικό λόγο. Θέλω η δημοκρατία να γίνει πραγματικότητα και να μην παραμείνει λόγια. Η κυρία Ροδούλα ζήσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ και εγώ εκ μέρου τη ελληνική αντιπροσωπεία που βρίσκεται σήμερα εδώ και του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την κυρία Άσκ και τον κύριο Επίτροπο, τη Σουηδική Προεδρία και την διακοινοβουλευτική αυτή συνάντηση με τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ενό προγράμματο που φιλοδοξεί να βοηθήσει στην προστιθέμενη αξία που χρειάζεται να πάρουμε για την συνομοθέτηση για την αρχή τη επικουρικότητα των εθνικών κοινοβουλίων αλλά κυρίως στα θέματα που αφορούν στην ελευθερία στη δικαιοσύνη και στην ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. ήθελα να απευθυνθώ σε εσά κύριε Μπαρό και να εκφράσω τα συγχαρητήρια στην ευρωπαϊκή επιτροπή στο πρόσωπό σας για το προσχέδιο που καταρτήσατε ως βάση του προγράμματος της στοκχόλμης το οποίο κατά τη γνώμη μας καθρεπτίζει μια πραγματικότητα μια κατάσταση και παρέχει προτάσεις για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος που αποκαλούμε κοινό χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες αφού υπάρχει η σχετική γνώμη των επιτροπών της βουλής των ελλήνων. θέλω όμως να επισημάνω επειδή αναφερθήκατε και σήμερα εδώ στις πολιτικές που ε, έχουν να κάνουν με την ελευθερία της διακίνησης της διασφάλισης της ιδιωτικότητας με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων για την πολιτική της μετανάστευσης και του ασύλου που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και για τους κοινούς κανόνες που πρέπει να υπάρξουν θα ήθελα να δούμε το μεγάλο ζήτημα του μεταναστευτικού προβλήματος για τις συνολικές πολιτικές που πρέπει να υπάρξουν και που αυτές σαφώς θα πρέπει να ακολουθηθούν από πολιτικές που αφορούν στο σοφρονιστικό σύστημα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σήμερα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ε, σε κάθε χώρα και κυρίως με τις χώρες της παραμεθόριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Επιτροπή, να προωθήσει η Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ε, έτσι ώστε να έχουμε βελτίωση των συνθήκων κράτησης και να βρούμε λύση, να εξευρεθεί μια λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών. Βεβαίως δεν αισθάνομαι καλά όταν μιλούμε για φυλακές σε μια Ευρώπη του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας που είναι το βαρόμετρο της δικής της αν θέλετε ουτοπίας ουτοπίας όμως που πραγματώνει τα όνειρα των ευρωπαίων πολιτών. θα ήταν καλύτερα να μιλούμε για σχολεία για την αύξηση αν θέλετε άλλων υποδομών στα πλαίσια πάλι της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης αλλά ωστόσο μια πραγματικότητα που υπάρχει ορίζει τελικά και το ερώτημά μου αυτό. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σισόν από την Πολωνική Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αναφερόμαστε στην Ευρώπη σαν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ίσως είναι από τα πιο σημαντικά ιδιαίτερα όταν συζητάμε κρίσιμα προβλήματα όπως αυτό της παράνομης μετανάστευσης. Δεν είμαι ο μόνος ούτε ο πρώτος ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα σήμερα βέβαια, αλλά είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορώ να το αγνοήσω. Εγώ είμαι Πολωνός, έρχομαι από την λεγόμενη κεντροανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια εμπειρία, όπως ξέρετε, το σιδηρούν παραπέτασμα. Έχουμε βιώσει μια φρικτή εμπειρία η οποία μας χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και οι συμπολίτε μου ακριβώς επειδή έχουν βιώσει μια τέτοια φιαλτική κατάσταση γνωρίζουν τι σημαίνει να νιώθει κανείς αποκλεισμένος και τι γνωρίζουν όταν μιλάει κανείς για προστατευόμενα σύνορα κτλ. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση λοιπόν συνάδελφοι να οικοδομήσουμε ένα νέο τείχος το οποίο θα διαχωρίζει την Ευρώπη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μια Ευρώπη δήθεν στην οποία σεβόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη μια Ευρώπη των χωρών οι οποίες είναι ουσιαστικά κράτη χωρίς δίκαιο και όπου οι πολίτες δεν καταφέρνουν να βλέπουν τα δικαιώματά τους να αναγνωρίζονται και συστηματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τέτοια σχηματική άποψη. Θα πρέπει να δούμε ε, πολύ προσεκτικά το τι συμβαίνει και σε επίπεδο δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο υπενθυμίζει πλέον συστηματικά ναι. ότι το άρθρο 8 θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη για τον καθορισμό και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών ιδιαίτερα όταν έχουμε κυρίως να κάνουμε με διαδικασίες επαναπροώθησης, με διαδικασίες εκδίωξης των παρονόμων μεταναστών, κάτι το οποίο προκαλεί τραγικές καταστροφές σε επίπεδο προσωπικής ζωής και οικογενειακής ζωής. Αυτό είναι μια σαφέστατη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν αναφέρεται κανεί στις ελευθερίε, στις δημόσιες ελευθερίες, βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ανάμεσα στην ομολογία του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και στην αντίστοιχη του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Przypomnę chociażby orzeczenie Trybunału Strasburskiego w sprawie przeciwko ιδιαίτερα όταν γίνονται ακροάσεις μεταναστών στα δύο δικαστήρια, η ερμηνεία η οποία δίδεται στα νομοθετικά κείμενα είναι εντελώς διαφορετική. Όταν υπάρχουν επίσης ε, ε, μερικές φορές προκαλούνται από δικαστικές αποφάσεις έρευνες και επεμβάσεις ε, σε αρχεία και σε γραφεία δικηγόρων και νομικών παραγόντων, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το άρθρο 8 και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Κοράτσα Μπίλτ δεν ακούγεται. Sorry. Uh, I would like to join uh, the voice of my distinguished... Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες συγχαίροντας και εγώ τη Σουηδική Προεδρία για την πρωτοβουλία uh, του προγράμματος Στοκόλμης το οποίο θα υποστηρίξουμε θα ήθελα να υπογρανίσω την πραγματική αφοσίωση της κυρίας Μπέα Σάσκη η οποία παλεύει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεταφέρουμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι εμείς δεν θέλουμε μια Ευρώπη φρούριο, θέλουμε μια ελεύθερη Ευρώπη. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε εδώ λίγο είναι η στάση και οι αντιλήψεις οι οποίες κυριαρχούν. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας αποδίδει μια τεράστια ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε. Πρέπει να είμαστε πιο επικοδομητικοί στις διαθεσμικές μας, στις διοργανικές μας σχέσεις και να είμαστε υπεύθυνοι, ε, να λαμβάνουμε συναποφάσεις θα έλεγα, με υπεύθυνο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνεί με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις ε, οι οποίες γίνονται δεκτές στο Συμβούλιο μόνο και μόνο επειδή από την 1η Δεκεμβρίου θα είμαστε τμήμα των συνομοθετών. Μια τέτοια στάση είναι ε, απαράδεκτη από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λυπάμαι πρόεδρο που δεν είμαι διόλου ε, διπλωματική. Ο κ. Πεζέτεμπερκ μας είπε χθε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει και περιμένω τις ιδέες ε, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό πέραν της ΚΟΖΑΚ η κυρία Μπεατρή Σάσκα είπε ήδη ότι είναι δυνατόν να συνδυάσουμε τον σεβασμό των αξιών μας και την ακαιρεότητα και τον σεβασμό μάλλον της ακαιρεότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών με την πραγματική φροντίδα της ασφάλειας των συγκεκριμένων πολιτών. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πιο πραγματιστική, μια λιγότερο ιδεαλιστική αν θέλετε Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη χρήσιμη για τους πολίτες. Και να υπογραμμίσω την ορθότητα αυτού που είπε ο Σίμων Μπουσουτήλ. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης απαιτεί μια πενταετία και είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω και επιμέρους να το προωθήσουμε βράχη πρόθεσμα για να δείξουμε με συγκεκριμένο τρόπο ότι δεν συζητάμε μόνο ιδέες λαμπρές αλλά προσπαθούμε να πετύχουμε και πετυχαίνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλτ. Η ε, κυρία Μπίθ από την κάτω βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Μπίθ μάλλον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε από δύο μιλητές από την Ολλανδία και τη Φιλανδία και συμμερίζομαι την άποψή τους ότι η συμμετοχή της Ένωσης στη σύμβαση αυτή πρέπει επιτέλους να υπογραφτεί. Η διαφορά της νομολογίας μεταξύ της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της σύμβασης αυτής σημαίνει πολλές φορές ότι μερικοί έχουν το δικαίωμα επιλογής ανάλογα με το τι τους βολεύει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο παρέπεμψε θέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά πώς θα ερμηνεύσουν τα εθνικά δικαστήρια αποφάσεις του ενός και του άλλου. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε για να βρούμε απαντήσεις και σε τέτοια προβλήματα. Δεύτερο θέμα. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, του οποίου είμαι αναφανθών υπέρ. Πολλές φορές προσπαθούν οι εγκληματίες να διαφύγουν από μία χώρα στην άλλη, αλλά αν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη στις δικαστικές διαδικασίες από χώρα σε χώρα, τότε θα μειωθεί η αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου και του ευρωπαϊκού εντάλματος. Αν κάποιος καταδικάζεται σε μία χώρα για αδικήματα στα οποία δεν θα καταδικαζόταν σε άλλη χώρα, μειώνεται προφανώς η αξιοπιστία. Επομένως το ευρωπαϊκό ένταλμα δεν πρέπει να καταλήξει τελικά να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει γιατί εκ πρώτης όψεως ο κόσμος το υποστηρίζει. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι η χρήση του πρέπει πάντοτε να είναι αναλογική. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαρτίνες από την Ισπανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Σουηδή Υπουργό Ασκ για την τεράστια εργασία που επετέλεσε κατά τη Σουηδική Προεδρία και συγχαίρω και τον Επίτροπο Μπαρό διότι και η Κομισιόν δούλεψε πολύ καλά. Τα δύο μάλιστα έγγραφα μας επιτρέπουν να ελπίσουμε ότι ρόδινο θα είναι το μέλλον. Επίσης ευχαριστώ όλους τους σημερινούς εισηγητάς γιατί πιστεύουμε ότι με την εργασία τους θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματά τους και στη δική μας δουλειά. Τώρα, για θέματα ελευθερίας, πληροφόρησης, δικαιοσύνης, θα ήθελα να πω ότι Ο Σαρτόρι το έθεσε ήδη το πρόβλημα. Η θέληση Vox Populi, Vox Day. Είχε λοιπόν τονίσει τον κίνδυνο που εκπροσωπούν οι ζηλωτέ και γνωρίζουμε ότι μία από τις βάσεις από τα θεμέλια της Ευρώπης είναι ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στο θέμα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην Ισπανία, πριν από δέκα μέρε, συνεδρίασαν οι παγκόσμιε αρχέ, διάφορε εταιρείε και οργανισμού προστασία δεδομένων. Υπάρχει μεγάλη προσδοκία και ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ένα κοινό μέσο προστασία δεδομένων και να έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και διεθνείς κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια, πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται να δημιουργηθεί αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και δικαστική συνεργασία. Εγώ θα πήγαινα και πιο μακριά, εναρμόνιση του ποινικού δικαίου σε ορισμένα πολύ ε, συγκεκριμένα ε, θέματα και αξιόπινες πράξεις. Υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης ε, της ποινική δικαιοσύνης στην τρομοκρατία, ας πούμε. Υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης στη δίωξη του εμπορίου ανθρώπων. Κυρίως όταν έχουμε δουλεμπόρους και ε, σκοπούς ε, τελικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Μπορούμε σε αυτά τα θέματα να έχουμε εναρμόνιση στην προστασία της παιδικής ηλικίας από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Και τελειώνω. Θα πρέπει επίσης να ε, ενισχύσουμε την κουλτούρα της συνεργασίας, την νοοτροπία της συνεργασίας. Γίνεται λόγος για δίκτυα εισαγγελέων, για δίκτυα ε, δικαστών, ανταλλαγή εμπειριών. Εγώ θα επέμεινα εδώ σε δύο στοιχεία. Πρώτον, ενίσχυση και προώθηση το στοιχείο της αμοιβή συνδρομής όταν έχει εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη στα συστήματα ποινική δικονομία, στι εγγύησει, στην κράτηση, ε, στην ε, ενημέρωση. Και επίση θα πρέπει να έχουμε συνεργασία και συντονισμό περισσότερο και θα ήθελα να μάθω και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Προεδρίας για τη δυνατότητα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λουίς Μιγκουέλ Παρίσα Καστάνος από την ΟΚΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπώ εγώ την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε είναι συμβουλευτικό όργανο, μια συνέλευση που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολίτων. Και εργαζόμαστε για την ανάπτυξη Ευρώπης, ε, οι οργανώσεις των εργοδοτών, ε, τα συνδικάτα, οι αλείς, οι αγρότες, οι οργανώσεις καταναλωτών, δηλαδή το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Ε, την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια τα 340 μέλη μας εγκρίναμε δύο γνωμοδοτήσεις για τη Στοκχόλμη. Η πρώτη αφορά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι η ατζέντα της Στοκχόλμης δηλαδή και το δεύτερο είναι γνωμοδότηση δική μας, η ίδια Πρωτοβουλία έτσι ώστε στο μέλλον οι πολιτικές μετανάστευσης να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις που διέπουν και προστατεύουν τα δικαιώματα αυτά. Σε γενικές λοιπόν γραμμές θα σας έλεγα ότι για την ΟΚΕ έχει πολύ μεγάλη σημασία, θεμελιώδη σημασία ε, το πρόγραμμα της Στοχόλμης και ιδιαίτερα αυτό που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες Έχουμε ανάγκη να ανήκουμε σε μια κοινότητα που να προστατεύει σωστά και την ασφάλειά μας και την ε, ελευθερία μας. Γι' αυτό επιζητούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν θυσιάζουμε τις αξίες της ελευθερίας και του κράτους δικαίου στο βωμό της ασφάλειας, για παράδειγμα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δίνουμε, παραχωρούμε ήδη την πρώτη νίκη στους τρομοκράτες. Γιατί δεν είμαστε πλέον μέλη μιας κοινωνίας ελεύθερης, ανοιχτής και δημοκρατικής. Το τελευταίο μου σχόλιο αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση, στην οποία είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι και στρατευμένοι. Η ΟΚΕ επιθυμεί η Ευρώπη να έχει κοινή πολιτική με εναρμονισμένη νομοθεσία, έτσι ώστε η μετανάστευση να γίνεται μέσα από νόμιμους διάβλους, διαφανείς και ε, ελαστικούς, και οι μετανάστες να έχουν σωστή και δίκαιη μεταχείριση. Για μένα λοιπόν ήταν απογοήτευση το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εγκρίνει η Σουηδική Προεδρία στο Συμβούλιο την οδηγία πλαίσιο για τα δικαιώματα των μεταναστών. Ελπίζω να το πράξει η Ισπανική Προεδρία. Και θα τελειώσω με μία ερώτηση, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπαρόντι, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωρίζει διότι συμμετέχει και είναι και συναρμόδιος μαζί μας για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ της ενσωμάτωσης, της ένταξης. Την περασμένη εβδομάδα συνεδριάσαμε με συμμετοχή όλων των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν τους μετανάστες στην Ευρώπη και υπερασπίζονται και τα δικαιώματά τους. Για συνεργαστούμε προς την ενσωμάτωση, την ένταξη των μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Ακριβώς από αυτή την άποψη της ένταξης των μεταναστών νομίζω ότι είναι λάθος μήνυμα να διαιρούμε το χαρτοφυλάκιο στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πρότεινε ο πρόεδρος Μπαρός. Διότι το να συνδέει τη μετανάστευση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι σφάλμα. Δηλαδή από κατασκευής, από την έννοια που συνδέεται η μία με την άλλη. Αυτό έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα, έχει κάνει με καταπολέμηση διακρίσεων η μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, παρακαλώ, από τη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στη χάραξη των πολιτικών για τον τομέα ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια που έως και σήμερα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κυβερνήσεων είναι μια ευκαιρία μια ευκαιρία για να ανακτήσουμε τη χαμένη ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ελευθερία γιατί τα τελευταία χρόνια στο όνομα της εξασφάλισης μεγαλύτερης ασφάλειας υποχώρησε πάρα πολύ το κράτος δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων χωρίς οι κοινωνίες μας να γίνουν ασφαλέστερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια έκανε βήματα αμερικανοποίησης και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι παράδειγμα ασφάλειας προς μίμηση. Είναι χρήσιμο στο τέλος της συνάντησης να ακούσουμε τις απόψεις της κυρίας Σάσκ εκ μέρους του Συμβουλίου και του κυρίου Μπαρό εκ μέρους της Κομισιόν για ορισμένες κρίσιμες αντιφάσεις και ερωτήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κυρία Άσκη και κύριε Μπαρό, πώς μας προτείνετε να έχουμε κοινέ πολιτικές σε αυτό το τομέα όταν οι κυβερνήσεις επέτρεψαν ένα απαράδεκτο opt-out στη νομική δεσμευτικότητα του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τρεις χώρες το ηνωμένο βασίλειο την τσεχία και την πολωνία. δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια μαύρη τρύπα μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεύτερον χρειάζεται περισσότερη συνεργασία των δικαστών και των αστυνομιών στην καταπολέμηση του εγκλήματος αλλά πώς θα νομιμοποιηθεί αυτή η συνεργασία αν δεν ισχυροποιήσουμε τους πολιτικούς ελέγχους πάνω σε αυτές τις εξουσίες έτσι ώστε να μην φοβάται ο κάθε πολίτης ότι στο όνομα της καταπολέμησης του εγκλήματος θα παρακολουθείται η ζωή του από το μεγάλο αδελφό και θα ήθελα σε αυτό το θέμα οι συνάδελφοι από την κεντρική και ανατολική ευρώπη να μην θέλουν να εφαρμόσουμε εμπειρίες που τις υπέστησαν και αυτοί από μια άλλη αυθαίρετη εξουσία. Τέλος, για τα θέματα της μετανάστευσης. Υπάρχει μια βασική αρχή στον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει στα χαρτιά, δεν υπάρχει στην πράξη. Η αλληλεγγύη το θέμα της μετανάστευσης όπως σωστά είπε και ο προηγούμενος ομιλητής δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μετανάστες είναι μια αδύνατη κοινωνική κατηγορία που δεν γνωρίζει καν τα δικαιώματά της. αντί λοιπόν να τα συρρυκνώνουμε στο όνομα της ασφάλειας πρέπει να τα ενισχύσουμε και να τους ενημερώσουμε και αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να τηρούμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου του ευρωπαϊκού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πράγμα που δεν κάνουμε. ένα τελευταίο για τον κύριο Μπαρό που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. κύριε Μπαρό, γιατί η ελλάδα η ισπανία οι χώρες εισόδου που δέχονται ένα μεγάλο κύμα μεταναστευτικής ροής να πληρώνουν μόνες τους το κόστος για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και γιατί πέρα από την οικονομική ενίσχυση να μην εγκαθιδρυθεί και μια δίκαιη κατανομή του κόστους στη στήριξη των μεταναστών που έρχονται εδώ. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία πλευρά ότι θέλουμε χέρια και μυαλά τα επόμενα χρόνια για να δουλέψει η ευρωπαϊκή οικονομία, να τους στέλνουμε αυτούς τους ανθρώπους ως εργαζόμενους και να μην τους αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Ευχαριστώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην πρώτη ολομέλεια τόνισα ότι θα πρέπει να ισχύσει ε, εγγύηση ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Τώρα θέλω να μιλήσω για την ελευθερία έκφρασης. Ορισμένα κράτη-μέλη και στο εσωτερικό της Ένωσης δεν σέβονται πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ μιλώ ως ε, μέλος ενός κόμματος που διαδέχτηκε ε, ένα κόμμα το οποίο απαγορεύτηκε το οποίο είχε όμως από το 15 μέχρι το 24% των ψήφων. Τι σημαίνει αυτό. Ε, γιατί το κάνει, γιατί μας απαγόρευσαν, γιατί τολμήσαμε να αμφισβητήσουμε ε, το δόγμα της πολιτισμικής κοινωνίας. Εμάς θέλουν, ε, τώρα μας διώκουν και με τα δικαστήρια να μας απαγορεύσουν και την ύπαρξη και τη χρηματοδότηση και να μας απαγορεύσουν το κόμμα μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ότι η Φλάνδρα είναι ένα έθνος εν το γεννάστε και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι η Ευρώπη των εθνών και των λαών. Και αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεν ακούμε αρκετά πράγματα γι' αυτό σήμερα. Και αυτό πρέπει να σας πω για την ελευθερία της έκφρασης, για τους εκπροσώπους ε, λαών ε, χωρίς κράτη και εθνών χωρίς κράτη. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στο Βέλγιο συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Και μπορεί αύριο να αφορούν το δικό σας κόμμα όλοι εσείς που κάθεστε εδώ. Ε, να ισχύσει λοιπόν η ελευθερία της έκφρασης και στο Βέλγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να διαπιστώσω εδώ ότι το πρόγραμμα της Οχόλμης το θεωρώ καταπληκτική και φανταστική μεταξέλιξη του παλαιού προγράμματος Τάμπερε και κατόπιν της Χάγης. Και βεβαίως συνδέεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας και είναι πραγματικό ποιοτικό βήμα ε, προς τα εμπρός στην Ευρώπη. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά και τα καλωσορίζω. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε κοινέ απαντήσεις για το άσυλο, για τη μετανάστευση κοινέ απαντήσεις γενικά, επαναλαμβάνω, και μια στρατηγική ασφαλείας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα θέματα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας και δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε πολλές φορές. Κάτι άλλο που θέλω να διαπιστώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που δίνει την καλύτερη απάντηση προς το παρόν σε αυτή την πρόκληση και για όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές και να απευθυνθώ στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και να πω ότι όσο σημαντικά και να είναι αυτό που κάνουμε εδώ και να με βρίσκουν σύμφωνο, είναι ένα βήμα όμως. Και θα πρέπει να προσέξουμε, να προχωρούμε με μικρά βήματα και με απλές ρυθμίσεις, διότι ένα βήμα στην Ευρώπη σημαίνει πέντε βήματα για τα κρατη δεν έχουν τον ίδιο διασκελισμό και δεν θα πρέπει να, να παραφορτώνουμε τα κράτη-μέλη για να ε, προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά συστήματα και στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γιατί αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια και τις κρατικές μηχανές και τους κατατόπους υπαλλήλους που καλούνται να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Τώρα για την προστασία των δεδομένων με ενθάρρυνε πάρα πολύ αυτό που είπε ο κ. Μαρτίνες της Ισπανικής Αντιπροσωπείας ότι ε, εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή, αλλά για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να αναζητήσουμε και πάλι την ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας του ατόμου και της ασφάλειας του συνόλου ή ακόμα και τη ιδιωτική σφαίρα και τη γενική ασφάλεια. Και πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι η σημερινή νέα ή πολύ νέα γενεά μεγαλώνει σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο με το διαδίκτυο όπου έχουμε μνήμη δεδομένων και για μεμονωμένα άτομα, ε, αν συνδυαστούν όλα αυτά τα δεδομένα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορεί να δώσουν μια πάρα πολύ στρεβλή και αρνητική εικόνα. Και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και ε, για την προστασία ε, της αυτοδιάθεσης του καθενός σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για το άτομό του. Γιατί φαντάζεστε θα πρέπει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να λέγουμε ποιος θα διαβάζει αυτά τα δεδομένα. Αυτά ήταν ε, τα τελευταία σχόλια ε, από τα μέλη και παραδίδω τώρα την Προεδρία στο συνάδελφό μου κύριο Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ για την, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο προείδρευσες και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν. Ο κατάλογος των ομιλητών έχει λήξει, εξαντληθεί. Συμφωνείτε, συμφωνείτε ότι έχει εξαντληθεί. Δεν διαμαρτύρεται κανείς και καμία. Θα ζητήσω λοιπόν από την Υπουργό Δικαιοσύνη της Σουηδίας να λάβει το λόγο. Ορίστε κυρία μου, ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και σας ευχαριστώ όλους για όσα είπατε. Είναι βέβαια δύνατο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ούτε όμως θα επαναλάβω αυτά που είπα στην πρώτη μου παρέμβαση. Θα σχολιάσω πάντως μερικά από τα σημαντικότερα που άκουσα. Καταρχήν, για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι προσπάθειες αυτές δεν πρέπει υπόθηκε να εφαρμοστούν χωρίς σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Συμφωνούμε με αυτό. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε μια εξισορρόπηση των δύο. Η καταπολέμηση του εγκλήματος τελικά αυτό είναι ο συνδυασμός των δύο. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει βελτιωθεί σε σχέση με την πρώτη του μορφή. Ο εκπρόσωπος της τσεχικής δημοκρατίας είπε ότι δεν γίνονται πάντοτε σεβαστά αυτά που είχαν προβλεφθεί από το πρόγραμμα, πρόγραμμα της Χάγης Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να λαμβάνονται αποφάσεις, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να εφαρμόζονται και γι' αυτό ένα τμήμα του προγράμματος της Στοκχόλμης αφορά ακριβώς τη συνέχεια, την παρακολούθηση και την εφαρμογή. Πρέπει να επιδείξουμε πρακτικό πνεύμα πράγματι. Το προσέξαμε στο πρόγραμμα της Στοχόλμης γιατί θέλουμε να μπορεί να καταλάβει ο πολίτης τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Τώρα για την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στις πληροφορίες ημέν των δε. Αυτό είναι θέμα καθορισμού προτύπων και για τα δεδομένα του DNA και για την ποιότητα των εργαστηρίων. Πρέπει οι πληροφορίες που έχουμε να είναι αξιόπιστες προφανώς ότι το εργαστήριο είναι αξιόπιστο, ότι η πληροφορία δίνεται με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα δικαστήρια κλπ. Αυτό επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι λεπτομέρειες αν θέλουμε να έχει αποτέλεσμα η συνεργασία είναι πολύ σημαντικές. Μερικοί επίσης μίλησαν για την αστυνομική συνεργασία μεν αλλά όχι τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο το πρόγραμμα της ε, Στοκόλμης. Είναι απλώς μια ευκαιρία για καλύτερο συντονισμό των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων. Περισσότερη συνεργασία που είναι απαραίτητη και η Ευρωπόλ μπορεί να αποτελέσει το κέντρο της συνεργασίας αυτής. Συνεργασίας με αστυνομίες και εκτός των ευρωπαϊκών χωρών. Η Europol είναι κάτι που προστίθεται στις εθνικές προσπάθειες και στις εθνικές αστυνομίες. Δεν υποκαθιστά τις τοπικές προσπάθειες και δραστηριότητες. Οι χώρες μέλη πρόσεξαν είδα ότι και μέσω των διμερών συναντήσεων που είχαμε ότι το θέμα της ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μερικοί είπαν να μην υπάρξει ούτε Ευρωπαίος εισαγγελέας. Στο πρόγραμμα της Στοχόλμης λέμε ότι τρεις είναι οι εναλλακτικέ λύσεις ως προς την ε, συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωδίκ, Eurojust. δεν είναι ένας ο τρόπος ή ούτε είναι απαραίτητη η δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ακόμη δεν αποφασίσαμε ποιος θα ήταν ο καλύτερος από τους τρεις τρόπους. Πολλοί επίσης ανέφεραν ότι δεν θέλουν να δημιουργηθεί μια Ευρώπη φρούριο από όπου θα αποκλείονται ορισμένοι. Αυτό είναι κάτι με το οποίο είμαι σύμφωνη. Υπάρχουν όντως δυνάμεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ανησυχίες του κόσμου για τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια υποδοχής τους με τον καταλληλότερο τρόπο. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης αφιερώνεται πολύς χώρος στο θέμα αυτό. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέχρι το 2020 είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε και με μεταναστευτικά θέματα είναι διότι αν δεν το κάνουμε τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να αποκλείσουμε τους πάντες από την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας οργανωμένος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος ώστε όσοι έρχονται στην Ευρώπη για οποιονδήποτε λόγο να την χάνουν τις κατάλληλης υποδοχή με κάποιους κανόνες και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης τους. Εδώ υπάρχει δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης συνεννόησης. Το Frontex καμιά φορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζεται σαν διοκτική δύναμη, δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Είναι ένα εργαλείο στήριξης των εθνικών δυνάμεων επιτήρησης των συνόρων αλλά και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σωστά το Frontex. Πολλοί ζητούν να λειτουργήσει καλύτερα το Frontex αλλά δεν κάνουν καμία πρόταση. Στο πρόγραμμα της Στοκόλμης προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί να υπάρξουν και περιφερειακά γραφεία του Frontex δηλαδή. Είναι μια δυνατότητα αντιμετώπισης και αυτή. Η έλεγχη στα σύνορα θα έπρεπε να είναι καταρχήν θέμα των εθνικών αρχών, αλλά το Frontex προστίθεται σε αυτά, συμπληρώνει. Για την ευρωπαϊκή συνεργασία θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κάτι μία πρόσθετη αξία. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά σε ενωσιακό επίπεδο δηλαδή από ότι σε εθνικό. Στην χθεσινή και σημερινή σας συνάντηση λοιπόν καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ήταν πολύ χρήσιμα όσα ακούσαμε και φυσικά δεν έχει ακόμα λήξει η διαπραγμάτευση. Η συνάντηση με προσώπους της Κομισιόν και της Προεδρίας καθώς και με εκπροσώπους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην Ένωση είναι κάτι πολύ χρήσιμο γιατί το όραμά μας είναι κάτι που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο και να αποτελέσει κίνητρο για τον τρόπο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της δωροδοκίας και διαφθοράς και της επίλυσης γενικότερα των σημαντικών κοινωνικών τους προβλημάτων. Βέβαια δεν είναι πάντοτε εύκολο και απλό θέμα να συνεννοηθούν κράτη με τόσο διαφορετικά προβλήματα, αλλά τέτοιου είδους συναντήσεις όπως με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ώστε η Ευρώπη να μην ε, αφοφύγει να συζητήσει τα προβλήματα των γειτόνων της και δεύτερον διότι ο κύριος στόχος της συνεργασίας αυτής είναι ειρηνευτικός. Θυμόμαστε όλοι τους πρόσφατους, τις πρόσφατες σειράξεις εκεί και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει συντονισμός της νομοθεσίας γιατί μόνο έτσι μπορεί με πεπολιτισμένο τρόπο να λυθούν τα προβλήματα μεταξύ ανθρώπων. Ως συνάντηση λοιπόν είναι ιδιαίτερα καλό υπόδειγμα της δουλειάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω και το πρόγραμμα της Λισαβόνας να σας δώσει ένα είδος πηξίδας, ένα πλαίσιο, έναν μπούσουλα για να εφαρμοστούν επιτέλους οι προθέσεις που θα διατυπώσουμε το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ μου. Σας ευχαριστώ γιατί κάνατε και μία χρήσιμη περίληψη θα έλεγα των προβλημάτων και διευκρινίσατε και κάποιες αμφιβολίες που είχαμε για τη συζήτηση. Ο κύριος Ινιάσιο Κωσίδο Γουτιέρες από το Ισπανικό Κοινοβούλιο θα ήθελε να σχολιάσει κάτι στα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας 3. Συμφώνησα με τον συμπρόεδρο εδώ ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ελάχιστος χρόνος. Ένα λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε σα σας ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τα συμπεράσματα της τρίτης ομάδας εργασίας για την προστασία των πολιτών και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας. Στην πρώτη παράγραφο λέγουμε ότι δεν υπάρχει εσωτερική ε, σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα στη ζωή και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν είναι εντελώς σωστό. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο, αν θέλετε, δικαίωμα. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει εσωτερική αντίφαση ανάμεσα στην ασφάλεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Εφόσον και ο εισηγητής της ομάδας εργασίας 3 μπορεί να απαντήσει, να συμφωνήσει σε αυτό το οποίο θέσατε, τότε η πρόταση, αυτή η μικρή αλλαγή είναι μια καλή αλλαγή. Ποιος είναι η συγητής της ομάδας εργασίας 3. Καλώς θα το δούμε αυτό. Είναι καλή πρόταση, Πρόεδρε. Είναι πολύ λογική η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά ο εισηγητής είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ξέρετε βέβαια ότι ο εισηγητής είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο σε τέτοιες συζητήσεις και γι' αυτό περίμενα από τον εισηγητή να πει το ίδιο με αυτό που είπατε εσεί, Αλλά χωρί τον εισηγητή και με τη δική σας βοήθεια αυτή η προφανή αλλαγή γίνεται δεκτή. Μπορώ να ζητήσω παρακαλώ τώρα τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρό, να πάρει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρία Άσκ που ανέφερε τα περισσότερα από τα προβλήματα επαρκώς. Εγώ θα προσπαθήσω απλώς, αν και είναι δύσκολο, να δώσω και εγώ ορισμένα στοιχεία απάντησης. Η κυρία Νταβίντ Ήταν σημαντικά αυτά που είπε, αλλά πρέπει και εγώ να επιμείνω για την πολιτική μετανάστευση. Ε, θα επιμείνω και εγώ δηλαδή στο θέμα της Ευρώπης του ασύλου. Ο κύριος Μαρίνταρη επίσης θέλησε να πω μερικά λόγια για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης προβλέπεται εταιρική σχέση με τρίτες χώρες που συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη. Είναι όντως έτσι μια νέα προοπτική. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουσουτήλ που είπε ότι μετά την ε, υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς πρέπει τώρα να δημιουργηθεί ο χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης κλπ. Προς τον κύριο Χρόλιτς θα ήθελα να πω ότι βεβαίως το θέμα δεν είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αστυνομία. Το Frontex απλώς συντονίζει τις προσπάθειες των χαρών μελών. Και ή ο έλεγχος στα εθνικά σύνορα είναι θέμα των χωρών μελών. Δεν πρόκειται εδώ για να αγνοήσουμε την ε, επικορικότητα. Είναι μια πρόσθετη αξία η ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ το φίλο μου Ζάκα Λέν Μπενιστή που έθεσε ένα κέριο πρόβλημα δηλαδή. Η αστυνομική και δικαστική ποινική συνεργασία αν θέλουμε να επιτύχει πρέπει να υπάρχει μία δομή ανταλλαγών που να αφορά όλα τα στοιχεία και δεδομένα και ευχαριστώ τη Σουηδική Προεδρία που επέτρεψε ήδη ήδη τη, να συμπεριληφθούν ορισμένες ρήτρες της συνθήκης του Προύμ στη Συμφωνία της Στοκόλμης. Μετά κύριε Μπενιστή, με το ΒΙΣ και ΣΥΣ 2 θα προχωρήσουμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομιών. Ο κύριος Γορέγγι Ρωτόντο επέμεινε ιδιαίτερα σε θέμα αμοιβαίας, το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Πράγματι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό δικαστικό πνεύμα ώστε η δικαστική συνεργασία να καταλήξει σε αυτή την αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο κύριος Κοθίδο Φυσικά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αστυνομία, αλλά και δεν θέλουμε να γίνει μπούνκερ η Ευρώπη. Θέλουμε να υπάρξει καλύτερη χρήση των των εργαλείων. Το είπε και η Βεατρίκη Άσκ, καλύτερη χρήση της Ευρωάστα, της Ευρωδίκα για την αντιμετώπιση των απειλών που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα, αλλά όχι φυσικά υποκατάσταση των κρατών. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Σάση, διότι έχει δίκιο. Πρέπει η Ένωση να συνυπογράψει την διάσκεψη των, την συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί έτσι αυτό θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Ο κύριος Μπράουν διαμαρτυρήθηκε, μα εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθεί ένα υπερκράτος. Είπα ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν αφαιρεί τίποτε από την εθνική, την εμπλουτίζει αντίθετα. Κυρία Σιζή, επέμεινε για κάτι που και μένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, οι συνθήκες κράτησης. Είναι κάτι που η Ιταλική Προεδρία επίσης είχε θέσει. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ανταλλαγής πειραματικών σχεδίων εναλλακτικής κράτησης. Κυρία Σισό, αυτή επέμεινε για κάτι το πολύ σωστό δηλαδή, την σύγκληση των νομολογιών μεταξύ Στρασβούργου και Λουξεμβούργου. Είναι προφανές ότι αν εγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορέσουν να λειτουργήσουν πολύ πιο συνδυασμένα. Η κυρία, κυρία Μπίλτ, ευχαριστώ και εκείνη που επέμεινε για τον ρόλο της, ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό γιατί και εγώ ήμουν εθνικός βουλευτής πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι η γνώση των εθνικών βουλευτών είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Αυτοί γνωρίζουν τις τοπικές πραγματικότητες. Τελεία. Ο κύριος Μπέης. μας είπε ότι υπάρχει κίνδυνος ε, αντίφασης μεταξύ νομολογιών αλλά αυτό το είπαμε και πριν ότι πρέπει να συνδυαστούν. Έχετε δίκιο δε για το ευρωπαϊκό ένταλμα. Καλό είναι εάν χρησιμοποιηθεί σωστά με αναλογικότητα. Αν θέλουμε να λειτουργήσει. Επίσης ευχαριστώ την, Ευρωπαϊκή Σουηδική Προεδρία που έκανε την πρώτη φάση, δηλαδή, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση, δηλαδή τις ελάχιστες εγγυήσεις. να υπάρχει μετάφραση και διερμηνία στις δίκες. Μαρτίνες. Πράγματι έχετε δίκιο για τα σοβαρότερα εγκλήματα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των κατηγοριών. Όχι ευρωπαϊκό ποινικό δικαίωμα, όχι, όχι, Πώς το πάρον, όχι, Αλλά για τα βαρύτερα εγκλήματα, για τα ιδεχθέστερα να υπάρξει μια συγκλισούλα. Κύριος Παριζά, Καστάνος. Εξ ονόματος της ΟΚΕ είπε ότι είναι όντως πράγματι απαραίτητη μια τέτοια σύγκληση. Οι μετανάστες είπε είναι κάτι που εμπλουτίζει την Ευρώπη εφόσον έχουν ενταχθεί σωστά. Πράγματι. Για τα δε δικαιώματά τους γίνεται, συμβαίνει πρόοδος. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης κάτι θα λέει. Ο κύριος Παπαδημούλης. Μα προχωρούμε κύριε, ακόμη κι αν ορισμένοι θέλουν opting out, προχωρούμε. Δεν είναι θέμα δημιουργίας κάποιου Big Brother, είναι απλώς θέμα να εγγυηθούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κύριε Σόφ. δεν έχουμε άμεσες αρμοδιότητες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά τα εγκρίνουμε. Τέλος ο κύριος Βος, τον ευχαριστώ. Πρέπει όντως να λάβουμε υπόψη μας και τις τεχνολογικές προόδους ως προς την προστασία των δεδομένων και θα εγκρίνουμε και κατοχυρώσουμε τεχνολογίες μόνο εάν είναι συμβατές με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την ιδιωτική ζωή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Να αυτά. Ίσως να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά τις άκουσα όλες όπως και η Βεατρίκη Άσκ με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σχεδόν ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Πέντε με επτά λεπτά ακόμα όμως. Γιατί έχουμε κάποια θέματα να ανακοινώσουμε στο τέλος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τη Σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπείται εδώ από τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Περ Βέστερμπεργκ και την κυρία Άσκ Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε ευχαριστώ για την εξαιρετική παρουσίαση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε και να τους χειροκροτήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Μπαρό, ε, αρμόδιο επίτροπο για ε, θέματα δικαιοσύνης, εσωτερικών και ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτησή μα. πάρα πολύ κρίσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας αλλά και για το έργο σας. Uh, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο συμπρόεδρο για να κλείσει. Να κάνει τα σχόλια τα τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκληση είναι αυτό για μένα τώρα να κλείσω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές ζήτησαν δράση κατά τη διάρκεια του διημέρου των συζητήσεών μας. Ε, σημαντικά θέματα όπως η διακρίση, η ανταλλαγή στοιχείων, καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος ε, τονίστηκαν ιδιαίτερα η Σουηδή Υπουργό Δικαιοσύνη, κυρία Μπεατρή Άσκ, περιέγραψε τι μα περιμένει τι επόμενε εβδομάδε. Ακούγοντα τι παρεμβάσει σα, διαπιστώνουμε ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ο μελλοντικό χώρος δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Σημειώνω ότι είναι σημαντικά τα θέματα και περίπλοκα για την εφαρμογή του προγράμματος Σοκόλμη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πάντα ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις ε, για τα θέματα αυτά, όπως ακριβώς ε, αυτό το διήμερο στην κοινή ε, κοινοβουλευτική μας συνδιάσκεψη. Όπως σας είπα ήδη, είναι εταίροι χρήσιμοι και επικοδομητικοί τα εθνικά κοινοβούλια για να διαβεβαιώνουμε πάντα ότι περνάνε τα μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις ρεαλιστικές για να διευκολύνουμε τις επόμενες μελλοντικές διαδικασίες του προγράμματος Σοχόλμης. Για το λόγο αυτό λοιπόν η Σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάσκεψη των Προέδρων ε, των ε, Κοινοβουλίων ζήτησε νέα συνάντηση στις 11 και 12 ε, Δεκεμβρίου και στη συνέχεια 14 και 15 Μαΐου του 2010 για να δούμε πώς θα ενσαρκωθούν όλα αυτά στην κοινοβουλευτική πραγματικότητα, στην κοινοβουλευτική δράση θέλουμε να βρούμε μέσα και διαδικασίες να εντείνουμε την ανταλλαγή ενημέρωσης και τη βέλτιση των πρακτικών για να γίνεται έλεγχος των κοινοτικών θεμάτων αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση τέτοιων ε, αρχών και στην αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να βρούμε τα μέτρα και τις διαδικασίες για να έχουμε αποτελεσματική ε, συνεργασία και συντονισμό των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Όπως είπαμε και χτες, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να βρουν πώς θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν αυτό το χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Πώς θα ασκεί το κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αγαπητοί βουλευτές, το τελευταίο αυτό διήμερο Εντοπίσαμε ε, κάποια σημεία που σίγουρα θα ελέγξουν οι επιμέρους ειδικέ κοινοβουλευτικές επιτροπές. Για να υπάρχει αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος χρειάζεται διακοινοβουλευτική συνεργασία. Τέλος, ελπίζω ότι θα μελετήσετε ε, το πρόγραμμα της Οχώνης αυτό το πολιετές και θα το ελέγξετε σοβαρά στα κοινοβούλια. Η συνθήκη Λισαβόνας αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα αυτό. Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεγκ ε, για τη συμπροεδρία της συνεδρίασης και του εύχομαι και όπως και το πρόεδρο της Ισπανικής Βουλής καλή τύχη στην επόμενη ε, διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε κύριε Βέστερμπεργκ. Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση λέγοντας ότι το θέμα που συζητήσαμε έχει τρομερή σημασία για τους πολίτες ελευθερία, δικαιοσύνη, ασφάλεια έδωσαν την δυνατότητα να θέσουμε πάρα πολλά προβλήματα όπως την ασφάλεια των πολιτών, τα δικαιώματα των πολιτών, διαμεθοριακό έγκλημα, μεταναστευτικές πολιτικές, ανθρώπινα δικαιώματα, Frontex, ναρκωτικά, τρομοκρατία, διαφθορά, προστασία δεδομένων, προστασία ιδιωτικών στοιχείων. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Mm-hmm. Έχουμε πλέον τρία έγγραφα στη διάθεσή μας τα οποία είναι καρπός των ε, ομάδων εργασίας. Έχουμε δηλαδή μια σωστή βάση για να προχωρήσουμε με το πρόγραμμά μας και να ξεκινήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος στη Στοκόλμη το Δεκέμβριο όπως ακριβώς το προτείνει και η Σουηδική Προεδρία. Την πρόταση αυτή προφανώς και θα την υποστηρίξουμε ιδιαίτερα σε κάθε προσπάθεια την οποία κάνει με μεγάλη ταχύτητα γιατί πρέπει να ανταποκρινόμεθα στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών τάχιστα. Να πω κάτι επιπλέον εδώ. Αυτά που είπαμε είναι σημαντικά, αλλά έχω και εγώ κάποιες υποχρεώσεις, θα έλεγα, να ξεφύγω λίγο από αυτό το οποίο συζητήσαμε. Να μιλήσω λίγο για την συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου 2009. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε πετύχει δηλαδή, θα έχουμε πετύχει κάτι για το οποίο δώσαμε μεγάλες μάχες και σε εθνικό επίπεδο γιατί έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε τις ευρωπαϊκές νομοθετικές δραστηριότητες, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο στο παρελθόν και είναι μια καλή εποχή επίσης και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αποκτούμε περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι στο παρελθόν και αυτά τα γνωρίζετε καλά. Η συνεργασία όμως μεταξύ μας πρέπει να είναι πραγματικά καλή, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την καλή συνεργασία και θα ήθελα να σας ζητήσω να ε, σταθούμε ο ένας στη διάθεση του άλλου για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες Είμαστε έτοιμοι για αμοιβαία συνδρομή και από τις δύο πλευρές απαιτούνται περισσότερες επαφές. Οι πρώτες επαφές θα ξεκινήσουν τον μήνα Δεκέμβριο ανάμεσα στους γενικούς γραμματείς όλων των κοινοβουλίων, εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα υπάρξει συνάντηση μετά προέδρων από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώνεται από τη Σουηδική Προεδρία. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποια δίκτυα επικοινωνίας. Έχουμε στη διάθεσή μας και την ΚΟΖΑΚ η οποία πάντα είναι σε λειτουργία. Έχουμε τις κοινέ διακοινοβουλευτικές συναντήσεις σαν αυτήν εδώ. Η επόμενη διακοινοβουλευτική συνάντηση θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και ζητώ συγγνώμη που ξέχασα μια τόσο σημαντική χώρα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι επισκέφθηκα την Ισπανία πριν λίγες μέρες και ετοιμάζονται πάρα πολύ σοβαρά για την Προεδρία τους. Και θα υπάρξει και άλλη μια κοινή διακοινοβουλευτική στα μέσα του επόμενου χρόνου. Απαιτείται συνεργασία όμως και σε επίπεδο ε, ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών απαιτείται να υπάρχει διακοινοβουλευτική συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Προωθούμε λοιπόν την δικτύωσή μας, τη συνεργασία μας και μέσω του διαδικτύου. Είναι κάτι το πάρα πολύ ε, αποτελεσματικό για όλους. Δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε σε καμία περίπτωση την νομοθετική μας δραστηριότητα. Η προετοιμασία μας λοιπόν είναι απαραίτητη και πρέπει να πάει καλά. Θα μου επιτρέψετε τώρα στο τέλος πλέον της συζήτησής μας ότι ευχαριστώ τον κύριο Περ Βέστερμπεργκ προσωπικά για την αφοσίωσή του σε αυτή την προσπάθεια, για τη συμμετοχή του στη συνάντηση αυτή και για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προετοιμασία αυτής της συνάντησης. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει όπως είπα κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνήθως Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους συνάδελφοι για τις συζητήσεις, για τις ιδέες σας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας. η κοινοβουλευτική στήριξη στις βασικές ιδέες που διέπουν θα έλεγα και χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης της επαφής ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθημερινή επαφή με τους συμπολίτε μας και θα πρέπει να υποστηρίξουμε πάντα τα ευρωπαϊκά όργανα, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις σας έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε στα μέσα του επόμενου χρόνου. Okay.